Okay, right, we'll start. Right, good morning, everybody. Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα γίνει μια μικρή τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με τα δύο θέματα που αφορούν τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά αντίστροφα, δηλαδή Πρώτα θα συζητήσουμε την συζήτηση υπό τον Βολφ Κλίν για την έκθεση πρωτοβουλίας και μετά θα συζητήσουμε τις τροπολογίες για την τροποποίηση του κανονισμού. Γιατί δυστυχώς θα, καθυστερήσει λίγο ο Ζαν Γκοζές και έτσι συμφώνησα να αντιστρέψω τη σειρά των δύο αυτών εκθέσεων. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και όποιο ενδιαφέρεται για αυτού του οργανισμού αξιολόγηση φαντάζομαι ότι ούτω ή άλλω θα πρέπει να είναι εδώ αυτή την ώρα. Θα, θα δώσω λοιπόν στον Βόλφ το λόγο καταρχάς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο Ζων Πόγκοζε ήδη είχε καταστήσει σαφέ ότι η δουλειά του αυτή τη στιγμή ουσιαστικά περιορίζεται και επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι η νέα υποίδρυση οργάνωση, οργανισμός ΕΣΜΑ στην επιτήρηση των ε, οίκων αξιολόγησης θα μπορέσει με το σωστό τρόπο να λειτουργήσει και να δράσει. Και αυτά που αποφασίσαμε στο παρελθόν ε, θα μπορέσουν να τροποποιηθούν. Τώρα στη δική μου έκθεση πρωτοβουλίας ουσιώδη θέματα, θεμελιώδη θέματα τα οποία δεν καλύφθηκαν μέχρι σήμερα αλλά τα οποία πρέπει να καλυφθούν πρέπει να εξεταστούν. Και το κάνω αυτό, αυτή την εξέταση, με απόλυτη συνένεση και σε καλή συμφωνία και συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει υπόψη μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι να επανεπεξεργαστεί τον κανονισμό αυτό εκβάθρων και στην τελευταία Παρασκευή είχαμε και την διαδικασία διαβούλευσης με τη δημοσίευση πολλών θεμάτων που εισήχθησαν έτσι στη συζήτηση είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων λοιπόν αυτή. Δεν μπορώ κάποια έτοιμα συμπεράσματα να διατυπώσω και να παρουσιάσω. Απλά θέλω να καταδείξω τα σημεία εκείνα με τα οποία θα απασχοληθώ στην ουσιώδη έκθεση, επί της ουσίας στην έκθεσή μου. Πρώτα απ' όλα να δούμε αν αυτό το business model, το πρότυπο λειτουργίας των οργανώσεων είναι το μόνο λειτουργικό και δυνατό και το καλύτερο. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή και οι τρεις, και οργανισμοί έχουμε υπόψη τους τρεις μεγάλους οργανισμούς που εργάζονται με την αρχή ότι ο issuer, ο εκδότης, πληρώνει. Δηλαδή, ο παραγωγός, εκείνος που τα προϊόντα του πρέπει να αξιολογηθούν, πληρώνει της, ε, ε, του οίκου αξιολόγηση και επιλέγει του οίκου αξιολόγηση και ο ίδιος εξάλλου. Αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν να ήταν πάντα αυτή η αρχή που λειτουργούσε. Δεν ήταν όμως αυτή η αρχή που λειτουργούσε πάντα. Στο παρελθόν υπήρχε και η προσέγγιση ότι ο user, ο χρήστης τέτοιου είδους ε, αξιολογήσεις από οικού αξιολόγηση πληρώνει. Αυτό όμως άλλαξε με τη ροή του χρόνου και σήμερα η μόνιμη προσέγγιση είναι ότι οι εκδότες, η παραγωγή προϊόντων οικονομικών πληρώνουν για αυτή την αξιολόγηση. Το κυριότερο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι το ότι εμείς συνολικά είμαστε της άποψης ότι υπάρχει πολύ λίγος ανταγωνισμός. Έχουμε τρεις οίκους αξιολόγησης που δρούν παγκόσμια και μόνο αυτοί οι τρεις είναι παγκόσμιοι. Στον τοπικό και περιφερειακό τομέα έχουμε πολλές ε, τέτοιες οργανώσεις όμως και φαίνεται ότι στην ΕΣΜΑ το, του χρόνου, όχι την 1η Ιανουαρίου βέβαια του 2011, αλλά την 1η Ιουλίου 2011 θα έχουμε την καταχώρηση που θα ξεκινήσει των rating agencies και μέχρι 50 μέχρι σήμερα εθνικές τέτοιες, εθνικοί τέτοιοι οργανισμοί, περιφερειακά δρόντες οργανισμοί θα καταχωρηθούν, θα παρουσιαστούν ώστε τουλάχιστον να έχουν την άδεια διασυνοριακής δράσης από την ΕΣΜΑ Λοιπόν, με άλλα λόγια τι σημαίνει αυτό. Το ενδιαφέρον και συμφέρον κάποιων που εμπλέκονται στην αγορά δραστήρια με αυτόν τον τρόπο είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός σίγουρα. Και για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός φυσικά αυτό είναι το προς το συμφέρον κυρίως πώς να το πω, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ίδιας και του Ευρωκοινοβουλίου και de facto είχαμε εδώ, έχουμε ένα ολιγοπόλιο ή σχεδόν μια μονοπωλιακή κατάσταση μπροστά μας και αυτό πρέπει να αλλάξει και εμείς πιστεύουμε ότι δημιουργούνται περιττές δαπάνες, υψηλές δαπάνες με αυτή την κατάσταση για τους χρήστες. Και αυτό θέλουμε να το καταργήσουμε ως κατάσταση, να το ξεπεράσουμε. Πώς είναι δυνατόν τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε, πώς να το πω, μια ευρωπαϊκή οργάνωση που υπηρεσία που θα συγκροτηθεί. Ε, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε ακόμα πιο πέρα και να το ξαναδούμε ή να το αξιολογήσουμε. Είχα προτείνει να έχουμε ένα είδος ιδρύματος, ένα ίδρυμα όχι public agency, δημόσια οργάνωση, δημόσιος φορέας που θα συγκροτηθεί, που θα εξαρτάται από κάποιο κράτος ή κάποια κυβέρνηση, αλλά ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που πρέπει να συγκροτηθεί με βάση το δίκαιο ή τους κανονισμούς και κανόνες ε, για τα ιδρύματα. Αυτό θα απαιτούσε βέβαια αυτό το ίδρυμα να ξεκινήσει με ένα κεφάλαιο εκκίνησης και το ερώτημα τίθεται, από ποιον θα διατεθεί, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρο είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί αυτό το κεφάλαιο εκκίνηση για να είναι ανεξάρτητο, ανεξάρτητο αυτό το ίδρυμα και στου φορεί και στου ε, στους φορείς που θα δραστηριοποιούνται ε, για την εποπτεία, να μην εξαρτώνται από κάποιο δημόσιο φορέα, κάποιο κράτο, κυβέρνηση κτλ. Κατά πόσον ένα τέτοιο ίδρυμα θα τύχει αποδοχή από την αγορά και από του εμπλεκόμενου στην αγορά είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξαναδούμε από κοντά. Το άλλο θέμα είναι η προσέγγιση που επιλέγουν οι Αμερικανοί, οι ΗΠΑ στο Reform Bill, στο νόμο, μεταρρυθμιστικό νόμο και να δούμε αν αυτό δίνει κάποιες ε, πολλά υποσχόμενες προοπτικές για μας. Στα μεταδιαρθρωμένα προϊόντα να υπάρχει διπλή αξιολόγηση double rating και ο πρώτος οίκος αξιολόγησης που θα μπορεί να επιλεγεί από τον εκδότη issuer για ο δεύτερος, ε, η δεύτερη, ε, ο δεύτερος οίκος αξιολόγησης δεν πληρώνεται από τον issuer αλλά από μια υπηρεσία εποπτείας. Μια και έχουμε με αυτό το πρότυπο, αυτή η προσέγγιση, στο τέλος τέλος το μονοπόλιο ή το ολιγοπόλιο που υπάρχει δεν θα το ε, άλλαζε σε, βά, ε, σε βάθος. Μετά τίθεται το θέμα μήπως ε, ζητάμε υπερβολικά, γενικά υπερβολικές αξιολογήσεις. Το θέμα τίθεται για το public, για τον δημόσιο τομέα. Αν σκεφτούμε τα δημόσια δάνεια και πιστώσεις, στο παρελθόν δεν ήταν συνηθισμένη υπόθεση ένας οίκος αξιολόγησης να αξιολογεί αυτές τις διαδικασίες. Σήμερα όμως είναι κάτι το αυτονόητο αυτό και ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε πολλά κράτη, η πλειοψηφία νομίζω των κρατών δεν πληρώνουν καν για τέτοιου είδους αξιολόγηση η Δημοκρατία της Γαλλίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πληρώνουν για αυτές τις αξιολογήσεις. Αυτοί που πρέπει να πληρώνουν είναι τα μικρά κράτη, μικρότερα κράτη που χωρίς αυτή την αξιολόγηση από τους οίκους αξιολόγησης δεν έχουν πρόσβαση σε δάνεια πιστώσεις στο κεφάλαιο από την τραπεζική αγορά. Αυτό είναι κάτι το αρνητικό να πληρώνουν οι Εσθονοί, οι μικρότερες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν έτσι εδώ να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Γενικά τίθεται το ηνωμενο βασιλειο δεν πληρωνουν για αυτες τις αξιολογησεις αυτοι που πρεπει να πληρωνουν ειναι τα μικρα κρατη μικροτερα κρατη που χωρις αυτη την αξιολογηση απο τους οικους αξιολογησης δεν εχουν προσβαση σε δανεια πιστωσει στο κεφαλαιο απο την τραπεζικη αγορα αυτο ειναι κατι το αρνητικο να πληρωνουν οι εσθονοι οι μικροτερες χωρες θα πρεπει λοιπον ετσι εδω να περιοριστει αυτη η κατασταση γενικα τιθεται το ερωτημα η αξιολόγηση κινδύνων μήπως και από πλευρά των χρηστών δεν θα έπρεπε υπό δική τους ευθύνη και δική τους διαχείριση να διοργανώνεται. Σήμερα είναι δεδομένο ότι έχουμε ένα σύστημα όπου καταρχήν de facto οι υπηρεσίες αξιο... οίκοι αξιολόγησης έγιναν ένα είδος ε, αρχής που εκδίδει πιστοποιητικά, πιστοποιούσας αρχής τίθεται το ερώτημα, έτσι πρέπει να είναι. Αν σκεφτούμε ότι οι οίκοι αξιολόγηση μέχρι σήμερα το απορρίπτουν, δεσμευτικά να είναι υπεύθυνες, υπεύθυνοι οι οίκοι αξιολόγηση για αυτά τα οποία εκδίδουν ω πιστοποιητικά ή ε, ω αξιολογήσει. Και λένε ότι εκδίδουμε μία άποψη, μία μη δεσμευτική άποψη, μία γνώμη που δεν είναι δεσμευτική. Ο χρήστη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι λοιπόν υπεύθυνη αυτή η οίκοι αξιολόγηση για τι συνέπειε των απόψεών του. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ανεχθούμε πιστεύω εγώ και δεν μπορούμε να το δεχτούμε να υφίσταται έτσι. Πρέπει να εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα αν και με ποιο τρόπο η οίκη αξιολόγηση για αυτά τα οποία προτείνουν και αξιολογούν θα είναι υπεύθυνη. Και αυτό δίνει πιθανότατα και τη σοβαρότητα και την ποιότητα για αυτούς τους οίκους αξιολόγησης και θα την διασφαλίζει αυτή την ποιότητα και αντικειμενικότητα και θα διασφαλίζει ότι δεν θα αντιμετωπίζουν τον πειρασμό αυτές, αυτή η οίκη αξιολόγησης σε σύγκρουση αρμοδιοτήτων ή συμφερόντων να ψάχνουν να βρουν μόνο τη μεγαλύτερη κερδοφορία η λύση, η επίλυση όλων αυτών των θεμάτων και οι απαντήσεις σε ιδανική περίπτωση θα έπρεπε να είναι παγκοσμιοποιημένη. Η αξιολογηση ε, δρούν παγκόσμια, θα πρέπει παγκοσμιοποιημένα μια ρύθμιση να ισχύει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ξέρουμε ότι η αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος, το rating ή μια χώρας ή μιας ε, διαδικασίας ε, εφαρμόζεται διασυνοριακά και έχει ισχύ διασυνοριακά και εκτός Ευρώπη και αυτά τα οποία γίνονται στις ΗΠΑ συμβαίνουν και εδώ σε εμά για τους επενδυτές από πλευράς ε, κρίσεων και αξιολογήσεων. Πρέπει να βρούμε μια ενιαία αντιμετώπιση, ένα ενιαίο πλαίσιο. Οι Αμερικανοί όπως είπα στη μεταρρύθμιση τους reform υιοθέτησαν μια συγκεκριμένη ε, κατεύθυνση. Το αν εμείς θα είμαστε πρόθυμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσουμε αντίστοιχα τέτοια μέτρα και να ακολουθήσουμε τέτοιες κατευθύνσεις, αυτό θα το δείξει το μέλλον. Σίγουρα δεν είναι διασφαλισμένο και δεδομένο το τι θα γίνει. Τώρα, συνοψίζω. Είναι σίγουρο ότι έχουμε πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν κύρια ερωτήματα. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε αυτά τα πλαίσια. Δεύτερον, πώς να μην υπάρχει over-reliance, υπερβολική εξάρτηση από τέτοιου είδους αξιολογήσεις. Η διαχείριση κινδύνου από τους χρήστες να μπορεί να διασφαλίζεται με καλύτερο τρόπο. Και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε η οίκοι αξιολόγησης να μην είναι υπερβολικά ε, ε, υπηρεσίες πιστοποίησης. Πώς μπορούμε δηλαδή να υποχρεώσουμε τους να είναι υπεύθυνοι και να υπομίζονται τις ευθύνες ε, των αξιολογήσεών τους και την αποζημίωση μιας πιθανής ζημιάς. Πώς θα αξιολογείται μια τέτοια ζημιά, πώς θα σταθμίζεται, ποιες κυρώσεις θα πρέπει μετά στη συνέχεια να υιοθετούνται να εγκρίνονται και ποιε δυνατότητε υπάρχουν ώστε τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, α πω πέντε ετών καταρχήν, ένα πενταετέ διάστημα, εμεί στην Ευρώπη να δημιουργήσουμε κάτι σαν μια ε, ε, υπηρεσία υποπτία του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελε το λόγο κάποιος από τους σκιώδεις εισηγητές. Σβέν. Μάλιστα. Όταν έχουμε ένα γερμανόφωνο εισηγητή πρέπει κανείς να μιλάει και γερμανικά αν μπορεί. Χαιρετίζω πρώτα αυτά τα οποία παρουσίασε ο συνάδελφος ο Βόλφ. Παρόμοια ερωτήματα και θέματα με απασχολούν και εμένα. Καταρχήν το θέμα για την εξουσία, την ισχύ στην αγορά Ουσιαστικά έτσι πρέπει να το πούμε. Πρέπει σε μια αγορά να υπάρχει ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό που υποθέτει ότι ο αριθμό των εμπλεκόμενων και τα μερίδια του θα είναι περιορισμένα στην αγορά. Γιατί κατά τα άλλα μπορούν να ασκήσουν, αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πολύ μεγάλη εξουσία και ισχύ στην αγορά η ισχυροί. Και εδώ τίθενται και τα ερωτηματικά. Υπενθυμίζω το θέμα της καλής αξιολόγησης των ΗΠΑ που εξακολουθούσε να είναι καλή. Μετά από αυτά τα οποία συζητήσαμε χθε με τον κύριο Γιούνκερ δεν το κατανοώ πως μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Είχα αρκετές συναντήσεις με τις μεγάλες, ε, τους εκπροσώπους των μεγάλων οίκων ε, αξιολόγησης και δεν με έπεισαν με τις απαντήσεις τους. Και αυτό πρέπει να είναι έναυσμα να ρωτήσουμε πώς μια τέτοια δομή αγοράς μπορεί να είναι αηφόρος και πώς μπορεί να είναι αξιόπιστη. Τίθεται τώρα το ερώτημα πώς θα διασφαλίζουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό Δηλαδή περισσότερους εμπλεκόμενους στην αγορά με μικρότερη εξουσία, με μικρότερη ισχύ από πλευρά τους. Είχαμε πει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγηση. Είχαμε πει να υπάρχει κρατικός οίκος αξιολόγηση. Για όλα αυτά τίθενται για μένα το θέμα αρχής. Δεν είναι τόσο αν θα είναι ένα ολιγοπόλιο ευρωπαϊκό ή αμερικανικό. Εμένα με ενοχλεί το ότι υπάρχει ολιγοπόλιο, άσχετα αν είναι αμερικανικό ή ευρωπαϊκό. Και το θέμα αυτό δεν θα το ε, ε, επιλύαμε αν, δημιουργήσαμε, δημιουργούσαμε κάποιες ε, μη θετικέ δομές. Πρέπει σε ευρύτατο πλαίσιο να δούμε τι μπορεί να γίνει για τις δομές των αγορών για να θεραπεύσουμε τα δυνά. Επίσης πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν ιδιωτική εξουσία στις αγορές όταν υπάρχει και υποψία ότι συμφέροντα δημιουργούν κάποιες καταστάσεις να αντικατασταθεί μια τέτοια κατάσταση από μια κρατική πλέον εξουσία όπου θα φοβάται κανείς και θα έχει την υποψία ότι πολιτικά πλέον συμφέροντα θα ε, ρυθμίζουν τα πράγματα. Τρίτη λύση, να βρούμε την λύση του Ιδρύματος. Ένα Ίδρυμα να εισαχθεί και να δράσει. Και στο ερώτημα παράδειγμα το οποίο διατυπώσατε εσείς. Πώς θα μεριμνήσει κανείς οι αξιολογήσεις ενός τέτοιου νέου εμπλεκόμενου δράστη να ε, είναι αξιόπιστες και σοβαρές. Τίθεται το ερώτημα, μήπως ε, αξιολογούνται ιδιαίτερα αυτές οι αξιολογήσεις μια και σε τακτά διαστήματα τους, τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν ζητούνται τέτοιες αξιολογήσεις, ρυθμιστικές αξιολογήσεις θα πρέπει και αυτό το Ίδρυμα να εμπλέκεται και να αξιολογεί και να εκφράζει την άποψή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ίδρυμα μόνο του θα δρά, αλλά δειγματοληπτικά ή ίσως και με θέματα συγκυρίας όταν υπάρχει δράση άλλων ε, οίκων αξιολόγησης να μπορεί αυτό το Ίδρυμα μικρότερους εμπλεκόμενους στην αγορά να τους υποστηρίζει και να τους ε, τονώνει με τις δράσεις του, με την υποστήριξή του. Ξέρω ότι εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση. Θα το χαιρέτιζα αν παρενέβαινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας έλεγε ποια είναι η άποψή της. Αν μπορεί αυτό δηλαδή να το υποστηρίξει ως πρόταση στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με τα αμφισβητήσιμα τα οποία σημειώνονται σήμερα στην αγορά πρέπει να δράσουμε. Ένα πολύ ψηλό ποσοστό των ratings ε, καλύπτει τους εκδότες, ε, τους ε, δημιουργούς παραγόγων και προϊόντων στην αγορά. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα υγιής αγορά να πληρώνει ο μαθητής το δάσκαλό του ο οποίος θα τον βαθμολογεί μετά στη συνέχεια κιόλας και θα πληρώνει ο μαθητής τα σπασμένα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε την ευθύνη πρέπει οποιοδήποτε εμπλέκεται στην αγορά να υπομίζεται την ευθύνη. Όποιο θέλει να κερδοφορήσει, κερδοσκοπήσει για παράδειγμα και υπάρχει ζημιά τρίτου να είναι υπεύθυνο αυτό για αυτή τη δράση του και να ε, μπορεί να υπομιστεί τι ευθύνε του οικονομικά. Και ένα τελευταίο. Θα το χαιρέτιζα ιδιαίτερα αν είχαμε στενή επαφή με, και παρακολουθούσαμε εκ του σύνεγγυ τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Υπήρχε ευρύτερη συζήτηση και στην πρόταση εξάλλου εξακολουθεί να υπάρχει ένα παράθυρο για τη συνέχιση αυτής της συζήτησης. Και γι' αυτό θα το χαιρετούσα καταρχήν. Αν αφενός εξετάζαμε σε βάθος τι αποφάσισαν οι Αμερικανοί, τι απέρριψαν και δεν υιοθέτησαν, να δούμε αμφωτέρωθεν δηλαδή της, ε, την εξέλιξη ε, των, πραγμάτων και των θετικών και εκείνων που δεν ε, ευδοκίμησαν και να δούμε τι συμβαίνει. Χαίρομαι και προσβλέπω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι κατεπηγόντως αναγκαίο πιστεύω. Μετά από τη μεταβατική περίοδο από την εποπτεία στην ΕΣΜΑ να δούμε τα προβλήματα εποπτείας τη αγορά με σωστό τρόπο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, I've got... Σας ευχαριστώ. Άσλι. Καλύτερα πρώτα εσείς και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο τέλος δηλαδή θα μιλήσει ο Φάμπρεγκας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Πάντα έχει να μας πει πράγματα που προκαλούν τη σκέψη. Θέλουμε να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό. Ε, και συμφωνώ με το τελευταίο που είπατε, ότι το λιγότερο που θέλουμε είναι να έχουμε ένα οίκο ε, που θα τον ε, διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνει και τριπλές αξιολογήσεις επειδή αυτό μπορεί να είναι από πολιτικής πλευράς ε, θεμητό. Και αυτό θα πούμε ότι θα είναι το αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά ένα δημόσιο ίδρυμα που είπατε, είναι ενδιαφέρον, public foundation, αλλά πόσο χρήσιμο θα είναι κάτι τέτοιο. Αναρωτιέμαι, θα ήταν χρήσιμο ή όχι. Χρήσιμο θα ήταν μόνο εάν έδινε μία γνώμη που θα, ήταν, ε, θα λαμβανόταν υπόψη από τις αγορές. Άρα θα έπρεπε να είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αν τελικά γίνει ένα εργαλείο μέσω του οποίου επιβάλλονται κάποιες πολιτικές απόψεις στις αγορές, δεν θα ενδιαφέρεται κανείς να ακούσει τι έχει να πει αυτό το ίδρυμα. Θα ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι οποιοδήποτε κράτος ή οποιαδήποτε επιχείρηση δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει έναν οίκο αξιολόγησης, αλλά επιλέγει να το πράξει. Επιλέ... Διακόπτεται ο μιλητής. Επιλέγει, επαναλαμβάνω, για να έχει καλύτερη τιμή για τα προϊόντα του ή της. Δεν μπορεί κανείς να σταματήσει μια τράπεζα από το να εκδώσει ομόλογα, παραδείγματος χάρη. Διαρωτώ με λοιπόν κατά πόσον η λύση που προτείνεται θα βελτιώσει την κατάσταση ή μήπως τελικά θα την επιδεινώσει. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι το κεφάλαιο μπορεί να πάει οπουδήποτε στον κόσμο και αν εμείς κάνουμε την πλέον περίπλοκη ε, περιοχή για την ε, συλλογή πόρων ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμος θα πάει και το χρήμα μαζί του θα πάει στην Κίνα, την Ινδία και σε άλλα μέρη, οπότε θα γίνουμε φτωχότεροι. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο έχω να πω και στο Βόλφ και στους άλλους συναδέλφους είναι ας μην επιδεινώσουμε τα πράγματα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια πλήρη αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο των προτάσεών της. Δεν θα ήθελα η Κομισιόν, αν δει ένα πρόβλημα, να πει κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι κάτι και στο κάνουν. Δεν θέλω να γίνει αυτό γιατί το τελικό αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο από αυτό που έχουμε τώρα. Και νομίζω ότι η Κομισιόν ε, χρησιμοποιεί αυτό ως πρόσχημα για να κάνει διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι πάντοτε ευεργετικά. Προσοχή λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Τζανίνη. Ζητήσατε το λόγο. Ε, είπατε το όνομά μου, όχι το επιθετό μου, γι' αυτό δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κλίντσε για τις πρώτες παρατηρήσεις που έκαναν και που αποτελούν έναυσμα για μια συζήτηση που δίχως άλλο θα συνεχιστεί. Δίχως άλλο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα όσα θα διατυπωθούν και σε διεθνές επίπεδο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στις συζητήσεις των G20 θα συμπεριληφθεί και το θέμα της αξιολόγησης ως ένας Τυχείο που έχει κανονιστική αξία. Τα όσα θα συζητηθούν στην διεθνή σκηνή θα πρέπει να αποτελέσουν τροφή για σκέψη για όλους μας. Τα σημεία που ανέφερε ο συνάδελφος Κλίνς καθώς και άλλοι συνάδελφοι, ο κύριος Γκίγκλον για παράδειγμα, με πείθουν καταρχάς σε ό,τι αφορά τον πλουραλισμό, τον ανταγωνισμό, την, τον αγώνα κατά της συγκέντρωσης που στην ουσία αποτελεί τη βάση της πρωτοβουλίας μας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η αξιολόγηση των χρεών των κρατικών χρεών, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως έδειξαν τα όσα διεμήφθησαν τα τελευταία αυτά χρόνια. Πάρα πολύ συχνά επιφανειακές αξιολογήσεις ή εικασίες για αξιολογήσεις οι οποίες διαψεύστηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη συζήτηση τίθεται και το θέμα του ευρωπαϊκού οίκου αξιολότησης που θα πρέπει να τύχει ε, μια εξέταση από εμά. Όλα αυτά είναι στοιχεία που δίχως άλλο θα εξετάσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι με την καθοδήγηση του κυρίου Κλίν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ορισμένους κοινού προσανατολισμούς. Thank It's, uh, I apologize for not uh, Καταρχάς να πω ότι λυπούμε γιατί δεν ήμουν εδώ και δεν άκουσα την πρώτη παρέμβαση, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την ε, άποψη ε, που θα εκφράσει εκ μέρους της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τους οίκους ε, αξιολόγηση, πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα της περιβολικής εξάρτησης και ότι τελικά ουσιαστικά δεν ασκείται δέουσα επιμέλεια για την αξιολόγηση. Θα ήθελα να ρωτήσω για τον εισηγητή και την Κομισιόν. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πράσινη βίβλος που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα. Um, Ευχαριστώ. Η νομίζω ότι ήδη είπε κάτι που θα ήθελα και εγώ να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα βέβαια να ευχαριστήσω τον Βόλφ για την παρουσίασή του που ήταν κατά την άποψή μου πολύ ενδιαφέρουσα και φυσικά και συμφωνώ ότι είναι διεθνέ το πρόβλημα. Έτσι, θα πρέπει να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία η οποία γίνεται ε, ανά τον κόσμο, να συμμετέχουμε σε αυτόν τον προβληματισμό για να βρούμε, αν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι, μια καθολική, μια οικουμενική λύση. Και πράγματι, πολλές φορές ε, οι ρυθμίσεις, οι κανονισμοί ε, παίρνουν, θέλετε, όμοιρο στις ε, αξιολογήσεις αυτές και δεν ασκείται ιδέως σε επιμέλεια. Εμείς θέλουμε να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση με κάποιους άλλους κανονισμούς μετά την κρίση, που εκπονήσαμε, αυξάνοντας δηλαδή τις απαιτήσεις περιδέουσας επιμέλειας. Και νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να ε, δούμε ποιο αποτέλεσμα, ποιο είναι ο αντίκτυπος. θα πρέπει να δούμε τελικά και τι κάνουν εξολογήσεις ε, στις άλλες ρυθμίσεις, στους άλλους κανονισμούς. Δεν μπορούμε να επαναχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα από τη θέση που έχουμε, αλλά γιατί να μην την εξετάσουμε και να δούμε αν είναι σωστά όλα τα μέτρα και διατάξεις και αν είναι και αποτελεσματικές. Τώρα για δημόσιο οργανισμό δεν νομίζω ότι θα ήμουν υπέρ και ακούστηκαν οι λόγοι από τους συναδέλφους. Κυρίως γιατί θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πολιτική παρέμβαση. Και σίγουρα θα πρέπει να σωματωθούν μηχανισμοί για την αποτροπή άσκησης πιέσεων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Βόλφ, να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα σου ξαναδώσω το λόγο εσέν για να συνοψίσεις. Η Κομισιόν, η κυρία Φάμπρεγκας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας που συζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Γιατί συμφωνούμε με τα όσα είπε ο κ. Κλίν στην αρχή, ότι δηλαδή υπάρχουν ε, θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα θυγεί. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν την προηγούμενη Παρασκευή το έγγραφο δημοσίων διαβουλεύσεων, το οποίο θα είναι ανοιχτό μέχρι τις αρχές ε, Ιανουαρίου. Στο έγγραφο αυτό περιγράφουμε μερικά από τα προβλήματα που θα πρέπει να εξεταστούν και προτείνουμε μερικές ενδεχόμενες λύσεις. Είναι ευχάριστο ότι διαπιστώνουμε ότι τα ίδια προβλήματα που αναφέρουμε κι εμείς είναι τα ίδια με αυτά που ετέθησαν εδώ σε αυτή την αίθουσα. Θα ήθελα να πω ότι από πλευράς Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντική η διεθνής, η παγκόσμια πτυχή που ετέθη από μερικά από τα μέλη της Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, ότι ε, πολλά θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο G20, συνεπώς η συζήτηση και οι δυνατές λύσεις θα είναι ευθυγραμμισμένες με οποιαδήποτε λύση θα προταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, στο οποίο βεβαίως συμμετέχουμε όλοι μας. Όπως ανέφερε η Πρόεδρος, το θέμα της, του πόσο βασιζόμαστε στις εξωτερικές αξιολογήσεις θα αντιμετωπιστεί αυξάνοντας τη δέοντα επιμέλεια και αυτό είναι κάτι που περιγράφουμε και στο δικό μας έγγραφο. Συνεπώς υπάρχει το θέμα του ανταγωνισμού Μία από τις δυνατές λύσεις για την αύξηση του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το τομέα είναι η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Κλίντς. Αυτό είναι μία από τις δυνατότητες που εξετάζουμε αλλά εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες όπως για παράδειγμα το ενδεχόμενο της δημιουργίας μεταξύ ΜΜΕ γιατί όπως γνωρίζετε από πλευρά της Επιτροπής το θέμα της βελτίωσης της ένταξη ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το τομέα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μας απασχολούν επίσης θέματα που έχουν σχέση με την ευθύνη. τα θέματα της ευθύνη είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα θέματα αυτά εξετάζονται και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα επιθυμούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε προσεκτικά όλα αυτά τα ζητήματα. Το άλλο θέμα έχει σχέση με τη σύγκρουση συμφερόντων. Το μοντέλο ότι ο εκδότης πληρώνει. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα βεβαίως που ε, υποβάλλονται από την Επιτροπή σε αυτό το δημόσιο έγγραφο. Το πέμπτο στοιχείο έχει σχέση με την αξιολόγηση του χρέους από πλευράς ε, της Επιτροπής μετά από την κρίση του κρατικού χρέους φρέτο στην Άνοιξη Διατυπώθηκαν πάρα πολλές επικρίσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αξιολογήσεις ε, του κρατικού χρέους από τις, τους οίκους αξιολόγησης. Και ειδικά το πότε αποκαλύπτονται αυτές οι αξιολογήσεις. Εμείς προτείνουμε ορισμένα στοιχεία που θα συμβάλλουν στην αύξηση του ελέγχου και της διαφάνειας αυτών των αξιολογήσεων που αφορούν ιδιαίτερα το κρατικό χρέος. Θα ήθελα επίσης να πω, όπως αναφέρθηκε στην αρχή της συνεδρίασης, ότι η Επιτροπή έχει σκοπό να υποβάλει μια νέα νομοθετική πρόταση μέχρι το ε, μέσο της επόμενης χρονιάς. Βεβαίως ε, θα εξετάσουμε λεπτομερώς όλες ε, τις απόψεις και όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης και βεβαίως θα γίνει μια πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την πρότασή μας αυτή. Βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα κοιτάξουμε την, ε, τα τελικά αποτελέσματα αυτής τη συζήτησης ε, που διεξάγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συναδέλφους και τις παρεμβάσει τους. Δείχνει αυτό ότι αυτό το θέμα πραγματικά ενδιαφέρει πολλούς από εμά και μας κινητοποιεί και πιστεύω στην αξιολόγηση της κατάστασης δεν βρισκόμαστε τόσο, σε τόσο διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βρετανό συνάδελφο ότι το κεφάλαιο πάει εκεί όπου έχει τις καλύτερες δυνατότητες κερδοφορίας και σίγουρα δεν μπορεί να είναι σκόπιμη προσέγγιση να δημιουργήσουμε νέα γραφειοκρατικά βάρη και επιβαρύνσεις. Δεν είναι αυτός ο στόχος σίγουρα, όμως μπορούμε ελπίζω μέσω μιας επιτυχούς δράσης, νέας κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουμε. Μπορούμε να το πετύχουμε η Ευρώπη ως έδρα επενδύσεων να κερδίσει και να μην χάσει γιατί θα δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους επενδυτές και τις, και ε, αποφάσεις τους. Λόγω μεγαλύτερου ανταγωνισμού θα υπάρχει το αποτέλεσμα τη δουλειά των οίκων αξιολόγηση που θα το δείχνει αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά σωστό είναι και ότι πρέπει να δούμε τις ε, σωστές κατευθύνσεις παγκόσμια. Συμφωνώ με τον Σβέν και το τι κάνουν οι Αμερικανοί και ότι θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να εξετάσουμε πόσο απέχουμε ο ένας από τον άλλο και κατά πόσο μπορούμε να βρούμε μια χρυσή τομή. Διότι όλα αυτά τα οποία βρίσκονται στη μεταρρύθμιση, στην πρακτική εφαρμογή, θα αλλάξουν πάλι λόγω των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών και του αποτελέσματος που έχει οδηγήσει τώρα οι Ρεπουμπλικανοί να έχουν το πάνω χέρι. Κάτι διαφορετικό θα θέλουν. Και αυτό το οποίο έχει επιτευθεί ως νομοθέτημα και ισχύει από πλευράς του Πρόεδρου Ομπάμα θα ε, μετεξελιχθεί και θα έχουμε και θα πρέπει να δούμε και τα θέματα υποπτίας. Ξέρουμε εμείς από την πλευρά μας ότι μέσω αυτής της, πώς να το πω, νέας κατεύθυνσης, νέων προσανατολισμών και άλλων μέτρων που θα υιοθετήσουμε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι στον χρηματοοικονομικό τομέα δεν θα ε, μπορούν να ελαφρύνουν το έργο τους ε, με την χρήση οίκων αξιολόγησης χωρίς να είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι και χωρίς να υπομίζονται τις ευθύνες για τις συνέπειες. Αυτό δεν γίνεται. Σίγουρα αυτό πρέπει να είναι και μια δευτερεύουσα πτυχή της δουλειάς μας που πρέπει να διασφαλίσουμε. Σίγουρα θα πρέπει για τον τομέα να δούμε ότι ε, υπάρχουν προβλήματα για τον ανταγωνισμό. Αυτό το δείχνουν και συζητήσεις με εκπροσώπους ε, που δείχνουν ότι θα ήταν θετικό να είχαμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Η συγκρότηση μιας νέας υπηρεσίας αξιολόγησης διακόπτεται ο μιλητής από κινητό. Για, αυτή τη, για αυτόν τον οίκο αξιολόγησης έλεγα, συνεχίζει, ότι δηλαδή πολλά χρόνια δεν μπορεί κανείς να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο τίποτα και αυτό είναι κάτι αποτρεπτικό δηλαδή ότι, δεν, ότι θα τίθεται πρόβλημα οικονομικό. Γι' αυτό κατέληξα σε αυτή τη σκέψη του Ιδρύματος. Αλλά στην πρακτική εφαρμογή του πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αν αυτά όλα δώσουν φτερά στον ανταγωνισμό και, τα προ, και τον προάγουν και αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ε, συνενωμένο στην Ευρώπη όπου θα μπορεί να δρά για την αγορά, θα πρέπει να σκεφτούμε αν τουλάχιστον θα μπορούσαμε να δίναμε κίνητρα με τέτοιο τρόπο εκεί όπου είναι υποχρεωτική η οίκη αξιολόγηση να λέμε ένα από αυτού του οίκου αξιολόγηση πρέπει να είναι καινούριο. Δηλαδή οι τρει παγκόσμιε υπηρεσίε, ή οίκοι αξιολόγηση να μπορούν να δρουν αλλά να μπορεί να εμπλακεί και ένας νέο τον οποίο θα ε, δημιουργήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίε και ανάγκη δράσης να ακολουθηθούν, ακολουθηθούν κάποιες νέες κατευθύνσεις στην αγορά, για την αγορά αγορά. Νέοι μη Χαίρομαι και προσβλέπω στη συζήτηση με τους συναδέφους για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Λείπουν οι συγκητές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την ημερησία διάταξη. Uh, Jean -Paul is... Ο Ζαν Πολ δεν μπορεί δυστυχώς να έρθει και το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Ποδηματά. Η κυρία Ποδηματά δεν έχει έρθει ακόμα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να διακόψουμε. Μέχρι να έρθει, μέχρι τις 11. Νάτι, νάτι, νάτι, ήρθε η κυρία Ποδηματά. Ταυμάσια. Ωραία, Διακόπτουμε για πέντε λεπτά μέχρι να τακτοποιηθεί η κυρία Ποδηματάκη και μετά θα ξεκινήσουμε. Καθίστε και πάλι παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και την κυρία Αποδηματά που ήρθε λίγο νωρίτερα. Κάποιες φορές ε, διαταράσει τη ρουτίνα. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 10 της ημερήσιας ε, διάταξης, χρηματοδότηση της καινοτομίας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν υποδηματά, είναι η συγγήτρια. Έχει το λόγο, Άννη. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, να μείνω στις κεντρικές ιδέες και στο σκεπτικό με το οποίο προσεγγίζουμε ε, αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας για τους καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης επειδή ακριβώς αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, γύρω από το σχέδιο έκθεσης θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις και προσεγγίσεις. Ε, ένα πρώτο βασικό σημείο ε, είναι ότι η συζήτηση για την, για την καινοτόμο χρηματοδότηση στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο επίπεδο δεν πρέπει και δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να είναι μια συζήτηση που θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στην ανέβρεση νέων πόρων η συζήτηση για την ανέβρεση νέων πόρων που είναι ασφαλώς ε, σημαντική θα πρέπει να συνδέεται με τις συζητήσεις και με τη διαδικασία μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό είναι το πρώτο σημείο με τις συζητήσεις σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση επίσης στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ασφαλώς με τις συζητήσεις για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάκαμψης και ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο επίπεδο. Η βασική θέση λοιπόν με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα των καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης είναι να προκρίνουμε ακριβώς εκείνες τις προτάσεις που ανταποκρίνονται σε αυτό το διπλό ή και τριπλό διακύβευμα το δεύτερο σημείο, όπως ε, ίσως σας διαπιστώσατε όσοι έχετε δει το σχέδιο έκθεσης, είναι ότι το κύριο ε, βάρος το δίνουμε στη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και αυτό πιστεύω ότι συμφωνούμε ότι σε μια περίοδο που οι κρατικοί προϋπολογισμοί και οι φορολογούμενοι Ευρωπαίοι έχουν επομιστεί το βάρος μιας κρίσης που κατά γενική ομολογία νομίζω οφείλεται στις εγγενείς αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού τομέα η διατήρηση της εξαίρεσης φορολόγησης του τομέα αυτού δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να δικαιολογηθεί πλέον ε, κατά κανένα τρόπο. Θεωρώ σημαντικό, έστω και αν δεν καταλήγουμε πάντα στα ίδια συμπεράσματα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα πριν από λίγες μέρες αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για την προσαρμογή του φορολογικού συστήματος κατά τρόπο που θα επιτρέψει στο χρηματοπιστωτικό τομέα να συνεισφέρει κατά τρόπο δίκαιο και ουσιαστικό στη χρηματοδότηση των δημόσιων προϋπολογισμών. Ο πρώτος λόγος, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι η συμβολή στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και στη μείωση της αστάθειάς τους, καθώς και των επιβλαβών επιπτώσεων από την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων αλλά και ορισμένων επικίνδυνων δραστηριοτήτων ο δεύτερος λόγος είναι η συμβολή στη δημοσιονομική εξυγίανση και στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια βιώσιμη ανάπτυξη όπως ακριβώς προβλέπει η στρατηγική ευρώπη 2020 και ο τρίτος λόγος με δεδομένη την απαλλαγή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω της αξίας των συναλλαγών μπορεί να συμβάλλει στην αναλογικότερη συμμετοχή του τομέα στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. άρα λοιπόν η ίδια η επιτροπή καταγράφει τους βασικούς λόγους για τους οποίους η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι αναγκαία. εφόσον λοιπόν συμφωνούμε σε αυτό το σημείο το επόμενο βήμα κατά τη γνώμη μου είναι να συνδέσουμε αυτή τη συζήτηση για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με το γενικότερο στόχο μας που είναι να επαναφέρουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα στην κύρια και πρωταρχική του λειτουργία που είναι η χρηματοδότηση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας ε, και για να το πετύχουμε αυτό είναι δεδομένο ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα φρενάρουν που θα αποθαρρύνουν απόλυτα κερδοσκοπικές και χωρίς καμία προστιθέμενη αξία συναλλαγές όπως είναι υψηλή συχνότητα συναλλαγές που οδηγούν συχνά σε σημαντικούς συστημικούς κινδύνους. Είναι σαφές κατά τη γνώμη μου ότι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών απαντά με τον καλύτερο τρόπο σε αυτή την πρόκληση. Σε ό,τι αφορά την εμβέλεια μιας τέτοιας φορολόγησης, δεν υπάρχει αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι καμία αμφιβολία ότι η καλύτερη λύση και ο πρωταρχικός στόχος μας πρέπει να είναι η επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας σε σχέση με τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρέπει όμως νομίζω να συνυπολογίσουμε το προφανές, το γεγονός δηλαδή ότι μέχρι σήμερα οι συζητήσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του G20 <clears throat> κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να χαιρετήσω τις γενναίες και αποφασιστικές πρωτοβουλίες της βελγικής προεδρίας που έχει θέσει την προώθηση του φόρου επί συναλλαγών ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες προτείνοντας μάλιστα τη συγκρότηση μιας ειδικής ε, υψηλού επίπεδου ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις ε, στα τέλη του χρόνου. Στο επίπεδο λοιπόν του G20 όπως σας έλεγα και πριν δεν έχουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις και κατά τη γνώμη μου το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο να πιέσουμε ώστε να φτάσουμε στη θέσπιση ενός τέτοιου φόρου παγκοσμίω. Το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά παγκοσμίω πιστεύω ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αποκρούσουμε το δίλημα περί αναμονής των αποφάσεων άλλων μεγάλων εταίρων και να ανοίξουμε το δρόμο για μια διεθνή συμφωνία προχωρώντας καταρχήν σε μια απόφαση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο και με το σκεπτικό που σας παρουσίασα πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο όπως το έκανε και στην περίπτωση της προώθησης των νέων κανόνων εποπτείας και λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου καθυστερήσει στην εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων που την έχουμε ζητήσει ως ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ήδη από τον περασμένο μάρτιο στο πλαίσιο του σχετικού ψηφίσματος που υιοθετήσαμε να καλέσουμε λοιπόν την ευρωπαϊκή επιτροπή να προχωρήσει ε, στην υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων άμεσα. πιστεύω ότι έχουμε κάνει ήδη ένα σημαντικό βήμα με την υπερψήφιση της έκθεσης Μπέρες για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, όπου ε, στην παράγραφο 73, όπως γνωρίζετε, ζητείται η επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με τη μεγαλύτερη δυνατή βάση, ε, όπως ακριβώς αναφέρει η παράγραφος 73, αλλά εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δεν συμβεί ο φόρος αυτός ε, να επιβληθεί καταρχήν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βάση λοιπόν αυτής της θέσης, με το σχέδιο έκθεσης που έχετε στα χέρια σας, ε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, κατόπιν ασφαλώς μελέτης επιπτώσεων, που θα λαμβάνει υπόψη την ισότητα των όρων ανταγωνισμού. Στην έκθεση περιγράφουμε με λεπτομέρειε ποιε θα πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μα οι βασικές παράμετροι ενός τέτοιου ε, φόρου. Ε, θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε αυτά. Ε, δεν, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες αυτού του είδους, διότι υπάρχουν στο σχέδιο της έκθεσης. Θέλω να πω δύο λόγια για τις προτάσεις για συνεισφορά των τραπεζών και για τον φόρο επί των κερδών ή επί των δραστηριοτήτων ε, από χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις έχουν ασφαλώς μια προστιθέμενη αξία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, κυρίως ως προς αυτή τη διάσταση που σας έλεγα πριν, δηλαδή το ρυθμιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ε, αυτός ο φόρος. Υπ' αυτήν την έννοια ο φόρος ε, ο φόρος ε, επί των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων ή επί των κερδών των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών νομίζω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτικός αλλά συμπληρωματικός του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δύο λόγια για τα ευρωομόλογα. Ε, θέλω να εκφράσω την ε, μεγάλη μου ικανοποίηση που η συζήτηση ε, γύρω από την έκδοση ευρωομολόγων έχει ξανά επικαιροποιηθεί. Θεωρώ ότι τα ευρωομόλογα μπορούν να αποτελέσουν το νέο πυλώνα για τη στήριξη των δημόσιων οικονομικών αλλά και να αποτελέσουν μια βασική ασπίδα για την ε, θωράκιση του ευρώ απέναντι στις, ε, στις επιθέσεις. Θεωρώ ε, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι χθε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Γιούγκερ, τάχθηκε υπέρ μιας ενδελεχούς εξέτασης της δυνατότητας αυτής σε επίπεδο ευρω, ευρωομάδας, από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων. Γνωρίζω ασφαλώς και γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις σχετικά με τη σκοπιμότητα έκδοσης ε, ευρωπαϊκών ομολόγων. Νομίζω όμως ότι στη σημερινή συγκυρία ε, είναι αδύνατο να παραβλέψουμε, είναι δύσκολο να παραβλέψουμε το τριπλό όφελος που προσφέρει η έκδοση κοινών ευρωπαϊκών ε, ομολόγων που είναι πρώτα απ' όλα η επαναφορά του κόστους δανεισμού των κρατών μελών σε λογικά επίπεδα δεύτερον η σημαντική επιπρόσθετη ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων ε, και τρίτον η λειτουργία τους ως ασπίδα ως ασφαλιστική δικλίδα απέναντι στις ε, επιθέσεις των αγορών. θα ήθελα ε, σε αυτό το σημείο στη συζήτηση για τα ευρωομόλογα να βάλω και μία ακόμα διάσταση τη σημασία των ευρωμολόγων ως ε, καινοτόμου πηγής χρηματοδότησης σημαντικών ευρωπαϊκών έργων και υποδομών μια διάσταση που έχει ε, υπογραμμίσει και ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής ο κ. μπαρόζο και αρκετά μέλη του κολεγίου των, ε, των επιτρόπων. το γεγονός αυτό νομίζω ότι υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ανάγκη να αποτιμήσουμε πλήρως αυτή τη φάση την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών ομολόγων και να προχωρήσουμε σε εκείνες τις ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης, ο φόρος άνθρακα τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς και σε μεταγενέστερο στάδιο θα πρέπει να το δούμε στις εισαγωγές από τρίτες χώρες ο φόρος αυτός πιστεύω ότι ε, μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μέσο φορολογικής δικαιοσύνης στη βάση της αρχής ορυπαίνων πληρώνει αλλά και να συμβάλλει άμεσα στην εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων της ευρωπαϊκής ένωσης σε σχέση με την ε, κλιματική αλλαγή. τέλος ε, και κλείνω κυρία πρόεδρε υπάρχει βεβαίως μια μεγάλη συζήτηση ως προς τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων που θα προκύψουν από αυτά τα νέα καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης. Ε, υπάρχει μια μεγάλη διάσταση απόψεων ως προς την διαχείριση αυτών των εσόδων. Θέλω να σημειώσω την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό όπου η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα αναφέρεται ως δυναμική νέα πηγή κοινοτικών ε, εσόδων και τέλος ε, να τονίσω το προφανές ότι πρέπει ασφαλώς να γίνει μια μεγάλη συζήτηση ε, γύρω από αυτό το θέμα της διαχείρισης των εσόδων που θα προκύψουν. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια ελάχιστη συμφωνία την οποία θεωρώ επιβεβλημένη ίσως και αυτονόητη ότι αυτά τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ανταποκρίνονται στην προστιθέμενη αξία ε, για την οποία εξ αρχής σχεδιάζονται ε, θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη ε, ότι ένα σημαντικό μέρος από αυτά τα έσοδα θα πρέπει να διατεθούν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση κεντρικής σημασίας, στρατηγικής σημασίας έργων και πολιτικών της Ένωσης. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα βασικά σημεία της έκθεσης πρωτοβουλίας για, τις, ε, για τους καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης. Ε, περιμένω με ανυπομονησία τις σκέψη σας και τις προτάσεις σας ε, για να φτάσουμε σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση σε ένα, στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οι πιο πολλοί σκιώδεις έχουν ζητήσει τον λόγο. Επομένως, θα ξεκινήσουμε, κυρία Χύπνερ, πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, εκφράζω το θαυμασμό μου για την τεράστια δουλειά που έχει κάνει η κυρία Ποδηματά. Θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία σημεία και να εκφράσω και κάποιες αμφιβολίες που έχω για ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία τίθενται στην έκθεση. Το πρώτο, το πρώτο θέμα που θέλω να σχολιάσω και η κυρία Ποδηματά το σχολίασε επίσης διαμακρών, είναι η αξιολόγηση επιπτώσεων, το impact assessment που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι μάλλον μπορεί να κολλησιεργεί, μπορεί να μην κολλησιεργεί η Επιτροπή, δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την αξιολόγηση και από ό,τι κατάλαβα του χρόνου το Μάρτιο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Νιώθω λοιπόν ότι Ίσως είναι λίγο νωρίς να ε, πιέζουμε για αυτό το φορό επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που προτείνεται ε, στην έκθεση. Γιατί αν δεν έχουμε αυτή την έκθεση εξολόγηση επιπτώσεων μπορούμε ίσως να μιλάμε για ε, την διόρθωση των ανισορροπιών στην αγορά, την παραγωγή εσόδων με, με διάφορα εργαλεία. Αλλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι επί της ουσίας για τα αποτελέσματα που θα έχουν τα διάφορα αυτά εργαλεία στα λεγόμενα externalities. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα αυτήν την μελέτη εξολόγηση επιπτώσεων. Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω σχετίζεται με κάτι που επίσης ε, μας παρουσίασε η κυρία Ποδηματά. Πάντα για το φόρο αυτό των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο την επιθυμία της αυτινούς, ότι θα πρέπει να επιμείνουμε και να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόρος στο παγκόσμιο επίπεδο και θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ε, γίνει στις επόμενες συναντήσεις της ομάδας των 20 να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Αλλά ό,τι λέει ο Ζαν Τρισέ και άλλοι που ενέχονται σε αυτές τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις ε, αν ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά, μάλλον είναι λίγες οι πιθανότητες και αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία, δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να εισαχθεί αυτός ο φόρος ε, μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, κατά την άποψή μου, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τον κίνδυνο μετατόπισης ε, των οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο σημείο 8 της έκθεσης λέγεται ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν βιώσει αρνητικό αντίκτυπο από την εισαγωγή ε, του φόρου επί των συναλλαγών. Δεν είμαι απολύτως βέβαιη ότι η σουηδική εμπειρία είναι τόσο θετική. Ίσως ο Όλισμιτ θα μπορούσε να επεκταθεί πάνω σε αυτό. Αλλά αν δείτε επίσης τι έγινε και στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον ε, γνωστό αυτό φόρο, βλέπουμε ότι οι Βρετανικές επιχειρήσεις ε, μετεγκαταστάθηκαν στην Ιρλανδία με την, μετά την εισαγωγή του, του φόρου εκεί. Άρα θα πρέπει και εκεί, σε αυτό το σημείο να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Επίσης, ε, στην έκθεση, ο φόρος ε, χρηματοπιστών συναλλαγών παρουσιάζεται ως μέσο για τη διόρθωση των ανισορροπιών των αγορών αληθεύει ότι υπάρχει κάποια σχέση, κάποια σύνδεση με βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και κερδοσκοπία, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λίγο υπερβολικό να πούμε ότι συνδέονται οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις με την κερδοσκοπία. Διότι κάποιες φορές δεν ισχύει αυτό και η CDO αυτή, αυτό, αυτό το εργαλείο το οποίο ουσιαστικά πυροδότησε και την κρίση ε, είναι ένα προϊόν μακροπρόθεσμης επένδυσης. Αν δούμε επίσης ε, και τους ε, όγκους συναλλαγών, τα trading volumes μάλλον θα μειωθούν οι όγκοι αυτοί αν εισαχθεί αυτός ο φως των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και θα αυξηθεί και η διακύμανση των τιμών, κάτι που μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κερδοσκοπία. Υπάρχουν μία δηλαδή τα οποία είναι ασαφή και αυτά θα διευκρινιστούν μόνο με αυτή την έκθεση αξιολόγηση επιπτώσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το FAT, αυτόν τον φόρο των χρηματοστηριακών δραστηριοτήτων κτλ. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε και σε σχέση με τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ότι δεν πρέπει να ε, τα θεωρούμε το ίδιο πράγματι υπάρχει εξαίρεση από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Αν θα μπορούσε να είναι ένα υποκατάστατο ίσως ε, για τον ε, ΦΠΑ αυτό το, αυτός ο φόρος, ε, αν τον οργανώσουμε καλά, ναι, ίσως θα μπορούσε. πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να ορίσουμε την προστιθέμενη αξία από ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή ίδρυμα. θα πρέπει να δούμε πώς θα φορολογούνται τα οικονομικά έσοδα του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία οφείλονται από την εξαίρεση από το ΦΠΑ. Και έτσι ίσως διορθωθούν οι ατέλειες ε, της αγοράς. Υποστηρίζω δηλαδή την εισαγωγή ενό φόρου FAT και είμαι πιο πολύ πέρα αυτού του φόρου παρά του φόρου FTT επί των χρηματοπιστών δηλαδή συναλλαγών. Και το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω σχετίζεται με τα ευρωομόλογα. Όταν μιλάμε για ευρωομόλογα, πολλές φορές με κάποια πράγματα. Υπάρχουν τα Eurobonds και τα project bonds ή European bonds όπως ε, ε, λέγονται στην έκθεση. Για εμένα είναι δύο διαφορετικά μέσα αυτά και αν τους δίνουμε την ίδια ονομασία, Euro bonds, ευρωομόλογα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν παρανοήσεις, να μην γίνει κατανοητό περί τίνος ε, ομιλούμε σε κάθε περίπτωση. Θα έπρεπε λοιπόν ίσως να τα διακρίνουμε, γιατί έχουν διαφορετικό στόχο και διαφορετικό μηχανισμό. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ποδηματά για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ενδεχομένω δεν συμφωνώ με όλα τα σημεία. Το θέμα είναι ότι φαίνει στην επιφάνεια μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. Εγώ είμαι φιλοευρωπαϊστή. θεωρώ τον εαυτό μου φεντεραλιστή. Δεν είναι καλό όμως να λέγεται στη χώρα μου. Μπορώ όμω να το πω με άνεση εδώ. Παράλληλα όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι Όλοι οι Ευρωπαίοι δεν αγαπάνε την Ευρώπη όπως την αγαπάμε εμείς εδώ οι παρόντες σε αυτή την αίθουσα. Και βεβαίως θα πρέπει τα όσα λέμε και τα όσα κάνουμε να έχουν μια βάση νομιμότητας. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειψη αυτής της νομιμότητας αυτές τις μέρες τα έγγραφα και η ρητορική είναι ωραία πράγματα, αλλά δεν καταφέρνουν να λύσουν αυτό το θέμα. Τα αποτελέσματα θα καταφέρουν να βρουν μια λύση. Προέρχομαι από μια χώρα που πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι ευτυχής όταν φορολογείται. Πρέπει να πω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις μέρες μας όταν προσπαθούμε να προωθήσουμε την ιδέα των μη φόρων σε γενική φάση. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο επιλύει τα προβλήματά μας. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Θα ήθελα να διατυπώσω ορισμένες παρατηρήσεις. Στα εκτιμώντας, το ιτολογικό, έχω την εντύπωση ότι διατυπώ αποτυπώνεται η ιδέα ότι την κρίση την επέφερε ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό. Ο τομέας αυτός έχει πάρα πολλά προβλήματα, μπορούμε να το διαπιστώσουμε εύκολα. Υπάρχει το θέμα της ρύθμισης, το γνωρίζουμε. Παράλληλα όμως θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, χώρες και υπουργοί οικονομικών και βουλευτές που θα πρέπει να κοιτάξουν και να αναρωτηθούν τι κάναμε εμείς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το σημείο στο οποίο έχουν φτάσει οι χώρες μας και για την ταχύτητα με την οποία έφτασε σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε ένα σημείο από, από την ιδεολογική έκθεση. Η κυρία Χιμπνερ αναφέρθηκε στο FTT, στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό δίχως άλλο είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Δεν είναι ευαίσθητο μόνο γιατί έχουμε προβλήματα με τις αποφάσεις, το πώς θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις δηλαδή. Πιστεύω ότι είναι δική μας ευθύνη να θεωρήσουμε κατά πόσον αυτό θα είναι αποτελεσματικό και βεβαίως και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα πολύ αμφιβάλλω. Αν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, εντάξει. Η κυρία Ποδηματά αναφερόταν στην έκθεση της κυρίας Μπερέσα. Μόνο ότι βεβαίως έγινε ξεχωριστή ψηφοφορία Πιστεύω ότι μπορούμε να ακούσουμε και τα όσα έχει να μας πει ο κύριος Τρισέ. Θα πρέπει όμως να δούμε τι εμπειρίες είχαμε σε αυτό το τομέα. Η κυρία Κιούμπρα αναφέρθηκε στο σουηδικό κακό παράδειγμα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν και τόσο καλό, καταστροφικό ήταν μάλλον. Μερικοί από τους συναδέλφους λένε ότι δεν μπορείτε να αναφέρεστε στην Σουηδία, είναι μια μικρή βόρεια χώρα, εδώ μιλάμε για την Ευρώπη ολόκληρη, υπάρχουν διαφορές. Δίχως άλλο υπάρχουν αγορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι το 83 Ξεκινήσαμε και καταργήθηκε αυτό το σύστημα αργότερα. Δεν ήταν επιτυχές. Μερικοί από τους ε, σοσιαλδημοκράτες ε, συναδέλφους θα μπορούσαν να, να το επιβεβαιώσουν αυτό, τουλάχιστον οι Σουηδοί σοσιαλδημοκράτες. Το άλλο θέμα είναι Εδώ στην έκθεση γίνεται αναφορά σε όσα κερδίσαμε, στα χρήματα που κερδίσαμε. Ποιος δεν τα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Θα, γίνει, θα δοθούν για αναπτυξιακή βοήθεια, θα δοθούν για θέματα περιβαλλοντικά στην Ευρώπη ή απλά και μόνο θα τα πάρουμε από τα ταμεία των ε, Υπουργείων Οικονομικών γιατί η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα χρέος. Θα πρέπει να μας δοθεί μια απάντηση. Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια, τα ευρωμόλογα. Είχα την εντύπωση ότι συμφωνήσαμε ότι αυτό το πρόγραμμα υποδομών θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα ευρωομόλογα. Έτσι τα αποκαλέσαμε ευρωομόλογα. Είχα την εντύπωση ότι ήταν ε, ο συμβιβασμό στην έκθεση τη κυρία Μπερέ. Μήπω θα μπορούσε να το εξηγήσει και η ίδια. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι από αυτή την άποψη θα μπορούσε να ήταν χρήσιμα. Οι Γερμανοί συνάδελφοι, ειδικά από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχεί με την ιδέα των ευρωμολόγων. Η κυρία Ποδηματά είπε ότι αυτό θα σώσει το ευρώ. Ενώ υπάρχουν Γερμανοί συνάδελφοι που θα υποστηρίξουν το αντίθετο, ότι θα προκαλέσουν προβλήματα τα ευρωμόλογα. Δεν θα συμβάλλουν ε, που δεν είναι στη διάθεση του ευρώ. Ο φόρος επί του άνθρακα. Έχουμε στη χώρα μου ένα φόρο επί του άνθρακα και θα μπορούσε αυτό να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αλλά ο στόχος αυτού του φόρου είναι να μειωθούν οι εκπομπές δεν είναι μία βιώσιμη βάση φορολόγηση. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μία αλλαγή της συμπεριφοράς μας. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι ένας χρήσιμος, καλός φόρος. Αναρωτιέμαι όμως αν είναι βιώσιμος και πιστεύω ότι δεν είναι βιώσιμος. Έγινε μια αναφορά στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η κυρία είμαι ανέφερε στην έκθεσή τη που θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα αυτό ακριβώ το θέμα. Ο δικό μου προβληματισμός και αυτό που θα πρέπει να τονίσετε στην έκθεσή σας κυρία Ποδηματά είναι ότι θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στις χώρες σας. Ε, καταφέρουν να επιτύχουν το στόχο της ε, χιλιετίας ό,τι αφορά το ΑΕΠ. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε στο σημείο αυτό, αν το θέμα που τίθεται είναι η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Εγώ με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω τις απαντήσεις σας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 που αφορά τις χώρες οι οποίες εισήγαγαν σύστημα παρεμφερών φόρων όπως είπατε φόρων συναλλαγών. Θα ήθελα να πω τελειώνοντας κάτι που συνήθως δεν λέγεται στα πλαίσια μιας επιτροπής. Λέω, δεν είναι και τόσο κακό πράγμα η κερδοσκόπη. Η κερδοσκοπία δεν είναι κατά ανάγκη πάντοτε κακή. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η απόδοση των ε, συνταξιωτικών ταμείων θα πρέπει να είναι υψηλή. Δεν υποτίθεται ότι θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα όπου κανείς δεν τολμάει να κερδοσκοπήσει. Η κερδοσκοπία είναι χρήσιμη σε μια ελαστική και λειτουργική αγορά. Ευχαριστώ. Εγώ, εγώ θα πρέπει να μιλήσω τώρα εκ του Φιλίπ. Εντάξει, μετά, μετά. Σας ευχαριστώ. Αντίθετα προς τον κύριο Σμιτ δεν είμαι εγώ υπέρ του ομοσπονδιακού χαρακτήρα όμως αυτό δεν με παρακολεί να συμφωνήσω με πολλά από τα επιχειρήματα που παρουσίασε και τόνισε όπως και κάποιοι άλλοι προλαλήσαντες και εγώ έχω αμφιβολίες πρέπει να πω όσον αφορά το έγγραφο το οποίο συζητούμε σήμερα θα προσπαθήσω όμως με την δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια να εξηγήσω τι εννοώ σε σχέση με αυτά. Αυτό το έγγραφο συζητείται σε μια χρονική συγκυρία και στιγμή όπου τα κράτη-μέλη και οι αρχηγοί κρατών βιώνουν βαθύτατες ε, μεταρρυθμίσεις και αλλαγές ε, στα δημοσιονομικά τους και στα θέματα του προϋπολογισμού τους και υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας όταν αντιμετωπίζουν αυτό το ιδιαίτερα περίπλοκο φαινόμενο, ιδιαίτερα σύνθετο φαινόμενο το οποίο είναι η υπεργύρανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε και ταυτόχρονα και μείωση της γεννητικότητας ε, Όλα αυτά δημιουργούν τεράστιες πιέσεις στα δημοσιονομικά μας και στα θέματα των προϋπολογισμών μας. Κάποια όχι μόνο εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επένδυσαν πάρα πολλά κονδύλια στο να αντιμετωπίσουν τα θέματα χρέους, υπερχρέωσης. Αυτά τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν εκεί δεν είναι διαθέσιμα αλλού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να εξηγιανθούν και να τεθούν εντάξει τα δημοσιονομικά. Και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα, το πρόσφατο συμβούλιο, την σύνοδο κορυφής που είναι ένα έκδηλο παράδειγμα όλων αυτών, ότι δηλαδή θα υπάρχει πολύ λιγότερη προθυμία από πλευρά των κρατών μελών να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα και συζητούμε αυτό το έγγραφο υπό αυτή τη συγκυρία, απλά επειδή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρειάζονται αυτά τα πρόσθετα χρήματα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι στην παρέμβαση μου θεώρησα ότι θα εκπροσωπούσα μία μειοψηφική άποψη. Έχοντας ακούσει όμως τις απόψεις των συναδέλφων, δεν είναι πλέον άποψη της μειοψηφία αυτό. Θα ήθελα να είμαι με μεγαλύτερο τρόπο, πιο, με πιο συγκεκριμένο τρόπο να αναφερθώ. Γίνεται λόγος για ένα ε, νέο, ε, μία νέα πηγή ε, φόρων, ένα νέο τέλος ή φόρο. Όλα αυτά προς ποιο στόχο είναι πολύ σημαντικό στην εισαγωγή, στην θέσπιση νέων τέτοιων φορολογικών μέτρων να γνωρίζουμε για ποιο στόχο και για ποια χρήση θα χρησιμοποιηθούν δεν συμφωνώ με την γενική ε, διαπίστωση ότι χρειαζόμαστε νέα κονδύλια, νέους πόρους για να αντιμετωπίσουμε κλιματολογικές αλλαγές ή για να αντιμετωπίσουμε τους στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης του 2020. Αυτά είναι πολύ γενικόλογα και αφηρημένα θα έλεγα. Με άλλα λόγια, οι δικές μου προτάσεις, αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν είναι να ακολουθήσουν άλλες κατευθύνσεις για να πετύχουμε συγκεκριμένους πιο εξειδικευμένους στόχους. Ένας από τους στόχους των τροπολογιών στην σύνταξή του ήταν από πλευρά μου το ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νέους φόρους ε, και φορολογικές πηγές που θα καθιστούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο ανταγωνιστική ή και καθόλου ανταγωνιστική κιόλας. Πράγμα το οποίο από πλευρά του θα σήμαινε ότι πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαζόντουσαν να εγκαταλείψουν ως έδρα επιχειρήσεών τους στην Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί τεράστιες επιφυλάξεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπήρχε συνολική συμφωνία στην εισαγωγή και έγκριση αυτού του κειμένου για αυτών των διαπιστώσεων. Και σε σχέση με την προηγούμενη διαπίστωση, αυτό που χρειαζόμαστε είναι, χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη ε, μελέτη επιπτώσεων πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσουμε και να σταθμίσουμε με ένα ανεξάρτητο αντικειμενικό τρόπο ποιοι ευρωπαϊκοί φόροι ή ποια ωφέλη θα μπορούσαν να αντληθούν από την εισαγωγή νέων φόρων, τέτοιου είδους φόρων. Θα ήταν πολύ θετικό λοιπόν υπό την μελέτη βιωσιμότητας να feasibility study να δούμε αν η εισαγωγή αυτών και έγκριση αυτών των κειμένων είναι εφικτή. Κάνοντας λόγο για τον φόρο στις συναλλαγές το FTT ή τον ε, φόρο το τέλος επί της ε, έκκλησης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις σε σχέση με την εισαγωγή του FTT. Ευχαριστώ. Yeah. Sorry. Συγγνώμη, Μιλώ εξ ονόματο του Φίλιπ Λάμπερ που είναι ο σχεδόν συζητητή ε, για αυτή την έκθεση. Βρίσκεται ακόμα δυστυχώ στην Επιτροπή Ίντρα, γι' αυτό δεν μπορεί να παραστεί. Όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, νομίζω ότι θα πρέπει πρωτίστως να πούμε τι στόχο έχουν και γιατί τα συζητάμε. Εδώ συζητάμε δύο θέματα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα εξισορρόπησης του προπολογισμού μας. Και πολλές χώρες αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες για να το επιτύχουν στα πλαίσια των υπαρχωσών δομών. Υπάρχουν υπάρχει ένας ανταγωνισμός, παγκόσμιος ανταγωνισμός για τη φορολογία που σημαίνει ότι δεν μπορούν να φορολογηθούν ορισμένοι τύποι εισοδήματο. Και υπάρχουν και τρόποι διαφυγής. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Το θέμα δεν αφορά τους νέους φόρους, αλλά αφορά την αποτελεσματικότητα του, τρέ, του παρόντος ε, φορολογικού συστήματος. Εκτός από αυτό, οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν μετά από αυτή την κρίση η οποία πυροδότησε πολλά στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν θα πρέπει τα έσοδα να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των εθνικών προπολογισμών. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα και μετά το απόγευμα θα συζητήσουμε την άποψή μας ε, για την έκθεση της χρηματοδότησης ε, της ανάπτυξης. Αυτό όμω είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Ένα θέμα που συζητιέται σε διεθνές επίπεδο. Πιστεύω ότι η λογική είναι διαφορετική, αλλά το μέσο είναι το ίδιο. Όπως λέμε τα γερμανικά, θα πρέπει να κρατηθούμε διαρκώς σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα πρέπει πρέπει να δημιουργήσουμε νέους φόρους. Δεν θα πρέπει να σταματήσει σοβαρή αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι μερικά από αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν με βάση τη φιλελεύθερη αγορά και να προσπαθήσουμε να βρούμε για ποιους λόγους δεν μπορούμε να διορθώσουμε μερικά από τα προβληματικά σημεία στην αγορά. Αυτό δεν έχει σχέση με αριστερά, δεξιά, φόροι, μη φόροι. Είναι θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν σοβαρά όπως συζητήθηκαν στην έκθεση περικλήσεις. Αυτό καταρχάς. Νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες μέλη είναι μέλη της ομάδας καινοτόμου χρηματοδότηση για την Αναβέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Ισπανία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μέλη αυτής της ομάδας και συζητάν το εργαλ... τα εργαλεία αυτά τα οποία μας παρέθεσε η κυρία ε, Ποδηματά στην έκθεσή της. Συζητάνε όμως και άλλα θέματα. Και αν τα συζητάμε αυτά τα θέματα, πριν περάσω στους τομείς που ήδη αναφέρθηκαν εδώ, θα ήθελα επίσης να πω τα σημεία που θα πρέπει να έχουμε κατά νου και που ανήκουν σε αυτά τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης. Ο τόχο είναι η μείωση του κόστου συναλλαγών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οι μετανάστε κερδίζουν χρήματα στο εξωτερικό. Αν στέλνουν όμω τα χρήματα ε, στι πατρίδε του, χρειάζεται να καταβάλουν ένα πολύ μεγάλο τίμημα για αυτή τη συναλλαγή. Δεύτερο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα επίσης των φόρων. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν την αγορά πολλών ε, φαρμάκων για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ακόμα και οι αναπτυσσόμενες χώρες τα φορολογούν. Και αυτό γιατί πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της δικής μου, δεν καταφέρουν να το κάνουν και για το λόγο αυτό υπάρχει ένας αθέμητος ε, ανταγωνισμός. Το τρίτο είναι το θέμα της καταπολέμησης, της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Μερικές φορές είναι δύσκολο να γίνει και από τις χώρες μέλη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή να φορολογηθούν ορισμένες, ε, ε, ε ένα μέρος των εσόδων. Συνεπώς, η γραμματεία της ομάδας παράλληλα με τις χώρες μέλη στην Ευρώπη που παρέθεσα ήδη θα πρέπει να δουλέψουν από κοινού για να αντιμετωπίσουν θέματα που αφορούν το εμπόριο. Θα πρέπει να διαπιστώσουν ποιος επωφελείται από όλα αυτά θα πρέπει να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα, την νομιμοποίηση παράγω, ε, ε, παράνομων εσόδων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό για να κλείσουν όλοι οι οδοί διαφυγής, η αποφυγής των φόρων. Δυστυχώς, μετά την ψηφοφορία ε, στην Επιτροπή Κρίσης, Χάρη στην κοινή προσπάθεια επετεύχθη μια συμφωνία, υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα το θέμα που ετέθη ήταν σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε είναι να ιδεολογικοποιήσουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαίνεται αυτές αναγνωρίζουν μερικοί όλες τις μορφές οικονομικών, δημοσιονομικών συναλλαγών που δεν μπορούν να φορο... χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που δεν μπορούν να φορολογηθούν. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Νομίζω ότι σαν ομάδα πρασίνων, εμείς σαν ομάδα πρασίνων ε, δημοσιεύσαμε μία μελέτη που παραθέτουμε τις διάφορες αγορές συναλλαγών και αυτή είναι μια πολύ πιο σοβαρή δουλειά. Είναι ορισμένα θέματα που μας απασχολούν περισσότερο. Το θέμα, ας πούμε, της ε, εμπορίας των βασικών αγαθών. Σε άλλα μέρη του κόσμου θα μπορούσε η φορολόγηση να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί η φοροδιαφυγή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είμαι κατά της ιδέας του να ιδεολογικοποιηθεί αυτό το θέμα. Πιστεύω, και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω, η υπάρχει ένα θέμα που αφορά την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Η κυρία Κιούμπνερ το έθιξε αυτό το θέμα. Είναι η απαλλαγή από το ΦΠΑ και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά το δημοσιονομικό τομέα σε σχέση με τους άλλους τομείς της οικονομίας, με τους άλλους τομείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι άνθρωποι χρειάζεται να πληρώσουν το τίμημα της ε, ε, κρίσης. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διορθωθεί. Συγγνώμη όλοι, αλλά θα ε, ξέρω ότι σου δημιουργώ κάποιο προβληματισμό. Το θέμα αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε για να επιτευχθεί και πάλι η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Κατά συνέπεια θα ήθελα να αποφύγουμε αυτή η συζήτηση, να γίνει μια συζήτηση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, μεταξύ των υπέρμαχων και ε, αυτών που είναι κατά των φόρων. Τα προβλήματα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης το πώς θα κλείσουμε τις οδούς διαφυγής, πώς θα δημιουργήσουμε καινοτόμου τρόπους χρηματοδότησης. Αυτό χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους γιατί δεν έχουμε εξετάσει αυτές τις μεθόδους, γιατί θα πρέπει να υποφέρουν διαρκώς και ε, να υφίστανται τις επιπτώσεις της κρίσης. Uh, Αγαπητέ συνάδελφε, μπορώ να σας πω ότι θα γίνει μία ακρόαση ε, στις 10 Ιανουαρίου και σε το χρόνο θα ενημερωθείτε για το πώς ακριβώς θα ε, γίνουν τα πράγματα. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους ε, να μην υπερβαίνουν το χρόνο αγόρευσης. Θα πρέπει το θέμα αυτό να περάσει στην Επιτροπή και μετά στην κυρία Ποδηματά. Να δώσω τώρα το λόγο στους επόμενους που ζήτησαν το λόγο. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος εκτός από αυτούς που ανέφερα. Όχι. Μαλίν. Κατανοώ την ανάγκη να είμαστε σύντομοι, αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. Κατανοώ την ανάγκη να είμαστε σύντομοι, αλλά είναι ένα ζήτημα αυτό που πρέπει να τύχει εμβαθυμένη συζήτηση. Θέλω επίσης ε, να ευχαριστήσω την κυρία Ποδηματά για καινοτόμες σκέψεις ε, πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμής δεν ήταν καινοτόμα και δεν ήταν δημιουργική όσον αφορά τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Και είπα ότι ω τμήμα μια παγκόσμιοποιημένη προσέγγιση πρέπει να το δούμε. Αναμένουμε αυτή τη σε βάθο μελέτη επιπτώσεων. Δεν μπορούμε να λάβουμε κάποιε αποφάσει εν κενό, αλλά πρέπει να ε, μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες κρίσεις για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση ακόμα και για να εξεταστούν λόγοι για την εισαγωγή ενός τέτοιου φόρου συναλλαγών με οποιαδήποτε μορφή αποφασίσουμε ότι θα είναι αποτελεσματικό κάτι τέτοιο και σε σχέση με τις ε, ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν θα επιβαρύνει μόνο την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν καινοτόμε σκέψεις να έχουμε και γι' αυτό αυτό προσπαθεί να κάνει η κυρία Ποδήματα με καινοτόμο τρόπο να προβληματιστεί με πρωτοπόρο, προπομπόρο όλο να δραστηριοποιηθούμε και στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή, μια και είναι μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλίας, μπορούμε να σκεφτούμε και το ασύλληπτο προσπαθώντας να καινοτομήσουμε. Προσπαθώντας να δούμε αυτό και βλέποντας ε, στην, ε, στις, ε, στον τύπο του Ηνωμένου Βασιλείου λέγοντας ε, ότι σε σχέση με το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ ε, θα μπορούσε να εισαχθεί ένας τέτοιος φόρος, ότι δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να αντληθούν, ότι χρηματοοικονομικά τέτοια ε, ποσοστά του 0,005% θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ίσπραξη 26 δις. Και αυτά θα σήμαιναν ότι υπό τη δική μου άποψη και πρέπει να πω ειλικρινά στο συνάδελφο εκείνο το οποίο δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε συγκεκριμένα επίπεδα. Μπορούμε να δούμε διαφορετικά επίπεδα ίσπραξης για αντιμετώπιση διαφορετικών προβλημάτων. Δεν είναι καθορισμός τελικού ποσού. Αυτά αλλά πρέπει να τα δούμε σε μεγαλύτερο βάθος ούτως ή άλλως. Και αυτό το οποίο βρίσκω πολύ ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση που εξετάζουμε σήμερα είναι ότι επικεντρώνεται σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σμιτ. Γιατί πρέπει να το κάνουμε. Διότι έχουν προβλήματα οι χώρες μας να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα και πρέπει να καλυφθούν αυτά. Και ένα πράγμα το οποίο αναφέρεται και νομίζω ότι είναι σε έντιμη έρευνα είναι ότι δεν μπορούμε να βασίσουμε όμως την άποψη μας μόνο σε ένα στοιχείο. Λέει όμως ότι σε σχέση με την, ε, τον ευμετάβλητο χαρακτήρα των αγορών που δεν μπορούμε να τον ε, ε, τι θα είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε για να σταθεροποιηθούν κάποια πράγματα και όχι να αποσταθεροποιηθούν. Βασίζοντας τις απόψεις μας σε αυτά πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε αρκετή έρευνα για αυτά τα ζητήματα. Επίσης λόγω των αλλαγών και μεταβολών σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν είναι ουσιαστικά πιο πιο εύκολο για χώρες να εισαγάγουν μονομερώς ε, κάποιες ε, τέτοιες ε, πηγές άντλησης φόρων και θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει δυσχέρεια. Όμως θα μπορούσαν πανευρωπαϊκά να εισαχθούν τέτοια τέλη. Το λέω αυτό επειδή έχουμε μια έκθεση που πρέπει να εξετάσουμε και δεν έχουμε απλά και μόνο τις, ε, ε, την έκφραση απόψεων. Η κυρία, για την κυρία Χιμπνερ. δεν είναι αληθές το ότι πήγαν στην Ιρλανδία βρετανικές ε, εταιρείες λόγω κάποιων συγκεκριμένων ε, κερδών. Πρέπει να πούμε ότι οι εταιρείε, όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε επιλέγουν για διαφορετικούς λόγους άλλες χώρες ε, ως έδρα των επιχειρήσεών τους και πρέπει να το δούμε αυτό. Το άλλο σημείο για τον φόρο χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων ναι μεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αλλά δεν ασχολείται με το θα έλεγα ε, μη δεδηλωμένο ε, συντελεστή των συναλλαγών. Θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε και αν μπορούμε να δράσουμε με αυτόν τον τρόπο και σε χαμηλό επίπεδο αυτό πρέπει να δούμε ότι μπορεί να είναι επωφελές και για την οικονομία. Απλά λοιπόν κρουοκόδωνα κινδύνου να μην χρησιμοποιηθούν μόνο τα μονοπόλια ή κάποια μονομερή επιχειρήματα και να πούμε ότι θα πρέπει να δούμε ε, από, αρκετούς, από αρκετές πλευρές ε, τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά του FTT. Λέγοντας ε, αυτά τα πράγματα σε σχέση με αυτή την ε, φορολογία, ξέρουμε ότι δεν είναι το θέμα της εφαρμογής ΦΠΑ, διότι υπάρχουν δυσκολίες εδώ και Ξέρουμε ότι δεν προλυαίνεται το έδαφος με αυτόν τον τρόπο. Ένα FTT λοιπόν, η μια μορφή ε, φόρου συναλλαγών είναι ένας τρόπος να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν ε, να ε, συνεισφέρουν όσοι εμπλέκονται στις αγορές και για να ε, εξομαλυθούν τα πράγματα. Θα ήθελα να πω στον κύριο Σμιτ και άλλους ότι δεν μπορεί να λέει κανείς ότι δεν είναι υπεύθυνοι οι τραπεζίτες, διότι οι ίδιοι οι τραπεζίτες έχουν συνεισφέρει με αυτές τις ευθύνες τους. Το να λέτε ότι δεν είναι η ευθύνη του χρηματοοικονομικού τομέα, δεν μπορώ να κατανοήσω τη λογική που σας εμπνέει να χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα σε σχέση με την πρόκληση της ε, κρίσης. Το είπατε εσείς αυτό. Και γι' αυτό εφόσον το άκουσα με αυτόν τον τρόπο αντιδρώ αυτό το οποίο εμείς ε, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, επειδή απογοητεύομαι να ακούω τα ίδια επιχειρήματα επανειλημμένα και ενώ δεν υπάρχουν επιχειρήματα κατά να λέμε δεν μπορεί να επιβληθεί ένα τέτοιο φόρο. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε τι αποδείξει. Αν πρέπει να αναμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσω πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο για να υποβληθεί αυτή η μελέτη. Έχουμε δυναμικό εμεί και α χρησιμοποιήσουμε αυτό το δυναμικό που έχουμε εμεί και α χρησιμοποιήσουμε άλλε μελέτε που βρίσκονται διαθέσιμε και που λένε ότι είναι απόλυτα εφικτό να επιβληθεί ένα τέτοιο φόρο στι συναλλαγέ σχεδιαστεί με αποτελεσματικό τρόπο και να μπορέσει να καταλήξει στο να αποφύγουμε την επανάληψη της σουηδικής κατάστασης πραγμάτων και του αδιεξόδου. Υπάρχουν λοιπόν αποδείξεις, που, στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν το ότι μπορεί να επιβληθεί ένας τέτοιος φόρος συναλλαγών και να μην λέμε διαρκώς ότι δεν μπορεί να το κάνουμε. Και στο τέλος αν πει μια μελέτη επιπτώσεων ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε τότε εντάξει ας το δεχθούμε. Αλλά δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής από κάποιο ίδρυμα ή από κάποιο θεσμικό ευρωπαϊκό όργανο. Γι' αυτό λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Um, um, Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε με τα ευρωομόλογα. Νομίζω ότι είναι ηρωνικό ακριβώς ε, τη στιγμή που εξετάζουμε το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης που υποτίθεται θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα οικονομικά τους κάνουμε παρατηρήσεις και δηλώσεις για τα ευρωομόλογα χωρίς να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ότι τα ίδια τα ευρωομόλογα θα φέρουν κάποιους ηθικούς κινδύνους, άρα θα μειώσουν την ευθύνη των κρατών μελών για τη διαχείριση των προπολογισμών τους. Επίσης έχει συζητηθεί το θέμα των ομολόγων project bonds για έργα υποδομών και σε μια άλλη επιτροπή το συζητούμε. Σε διάφορες ε, περιοχές του κόσμου υπάρχουν, της Ευρώπη συγκεκριμένα, υπάρχουν ανάγκη για επενδύσεις και για έργα και για τι στόχους ε, της Ευρώπης 2020 και πέραν αυτού του χρονικού ορίου. Και επίση οι δημόσιε επενδύσει και οι ιδιωτικέ επενδύσει μπορούν να είναι ευεργετικέ. Θα πρέπει όμω ε, να υπάρχει κατάλληλη διαφάνεια, διαχείριση κινδύνων και να μην μιλάμε για χρηματοδότηση που ε, όπως και το δικό μου ε, κράτος μέλος ε, έφερε, στο δικό μου κράτος μέλος έφερε πολλά, πολλά προβλήματα. Θα πρέπει και για αυτά τα ομόλογα project bonds να υπάρχουν έλεγχοι. Κάποιοι είπαν ότι το κατάλληλο σημείο είναι η EIB, η Τράπεζα Επενδύσεων αλλά ε, δεν θα ήμουν απαραίτητα σύμφωνη με αυτό. Θα πρέπει να προσέξουμε και το εξή. Ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να βάλει χρήματα σε κάποιο έργο, αλλά μπορεί να μην είναι χρηματοδοτήσιμο αυτό το project, γιατί πάντοτε την πρώτη απώλεια την έχει ο δημόσιος τομέας ή το πρώτο κομμάτι το χρηματικό. Θα πρέπει να δούμε επίσης τις αρχές που θα πρέπει να ε, διέπουν τον προπολογισμό. Δεν θα πρέπει ε, να υπάρχει έλλειμμα και δεν θα πρέπει να βάλουμε έλλειμμα από την πίσω πόρτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ε, φόρους επί των συναλλαγών, πράγματι είναι ιρανικό και έχω ακούσει όλες αυτές τις συζητήσεις για την εποπτεία κτλ. Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο Σβέν, υποστηρίζουν ε, αυτά που λέει ο Τρισέ τελικά που μας προειδοποιεί και μία από τις πρώτες προειδοποιήσεις του ήταν «Σας παρακαλώ μην αναφέρετε μονομερώς στην Ευρώπη ένα φόρο πετών συναλλαγών». Δεν τον ακούνε όμως, δεν ακούνε αυτή την προειδοποίησή του. πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Βρετανική εμπειρία, η κυρία Χούμπνερ ε, μίλησε γι' αυτό, θέλω να πω ότι ναι, πράγματι ο επικεφαλής ε, του χρηματοστηρίου ε, του Αγγλικού μίλησε για αυτό το φόρο, stamp duty, φόρο χαρτοσύμου. Πράγματι έχει, ε, έχουν επικαλεστεί οι μεγάλοι παίκτες αυτό το φόρο. Τελικά οι μικροί επενδυτές τον πλήρωσαν, επομένως δεν ήταν και τίποτα το εξαιρετικό ως λύση. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις αδιαφανείς δεξαμενές, αυτές τις αγορές παραγόγων και όλα αυτή την αδιαφάνεια. Ίσως φαίνονται ωραίοι όλοι αυτοί οι φόροι, αλλά πρέπει να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ τον Σβέν για το σχόλιο που έκανε, ιδίως ό,τι αφορά την ε, αγορά ε, αγαθών. Επίσης, Όλεκ είπε ότι υπάρχουν κάποιοι ε, φόροι, οι οποίοι όμως δεν πρέπει να είναι μόνιμοι, αλλά να οδηγούν σε αλλαγές συμπεριφοράς και συμφωνώ. Υπάρχουν μεμονωμένοι φόροι άνθρακα όμως σε διάφορα κράτη-μέλη. Μήπως τελικά το να εισαγάγουμε έναν ενωσιακό φόρο άνθρακα, αυτό είναι σε βάρος των εθνικών φόρων άνθρακα που εφαρμόζουν ε, διάφορα κράτη-μέλη. Την Παρασκευή Ήμουν σε έναν ε, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο εμπορευματικό σταθμό ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχω δει, ε, είδα μάλλον, τεράστια και άδεια κοντέινερ από την Άπο Ανατολή, τα οποία μένουν στι αποθήκε εκεί και δεν πρόκειται να γυρίσουν ποτέ πίσω. Λοιπόν, πρέπει να φροντίσουμε να μην επιδεινώσουμε τα πράγματα, ακολουθώντα κάποιε συγκεκριμένε κατευθύνσει Και το τελευταίο που θέλω να πω Ίσως στη Γερμανία, γιατί ο Σβέν κάτι μου λέει, μπορεί να φεύγουν από τη Γερμανία, δεν ξέρω. Ε, σε εμά πάντως μένουν εκεί. Λοιπόν, το τελευταίο σημείο για την αύξηση των φόρων, χωρίς να λέμε πού δαπανούμε τα χρήματα. Φυσικά και τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξοικονομούν πόρους. Και σίγουρα θα πρέπει να εξηγούν καλύτερα και στην κοινή γνώμη πού πηγαίνουν οι αποταμιεύσεις. Σίγουρα είναι δύσκολο το να γίνουν αποταμιεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο μπορεί καλύτερα να κάνει επιχειρήσεις και να αποταμιεύει και ε, όχι μόνο να κοιτάμε τα θέματα καινοτόμου χρηματοδότησης. Ο Γκούναρ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση. Τρεις παρατηρήσεις θα είχα να κάνω. Πρώτον για τα ευρωμόλογα τα οποία πιστεύω και αναφέρθηκε αυτό, αντιβαίνουν αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Θα πρέπει να έχουμε κυρώσει τα ευρωομόλογα είναι εξουδετέρωση, μείωση, συρρήκνωση των, ε, των επιπτώσεων των κυρώσεων. Αλλά υπάρχει και άλλη ε, συνέπεια επίσης, διότι τα ευρωομόλογα και δεν κάνω λόγο γενικά, γενικόλογα, θα σήμαινε ότι οι πολίτες σε χώρες με υψηλότερους φόρους και εξισορροπημένους ε, ισολογισμούς και δημοσιονομικά θα πλήρωναν περισσότερους φόρους και θα επιβαρυνόντουσαν περισσότερο. Και αυτή είναι η συνέπεια δεν μπορώ να υπομισθώ την ευθύνη να επεξηγήσω όλα αυτά στους πολίτες εκείνων των χωρών με υψηλότερη φορολογία που πληρώνουν περισσότερου περισσότερους φόρους ήδη σήμερα για μια τέτοια κατάσταση. Δεύτερον, για τον φόρο τέλους έκκλησης διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει εξ ορισμού να προσπαθήσουμε να έχουμε έναν αϊφόρο, ε, ένα αϊφόρο τέλος. Και έτσι λοιπόν θα είναι περιορισμένη η διάρκεια αυτού του φόρου. Όμως οι διαφορές στις χώρες μας μας δίνουν ένα προφανή λόγο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο, διότι οι διαφορές μεταξύ Πολωνίας και Σουηδίας, για παράδειγμα, είναι τεράστιες και οι επιπτώσεις μπορώ να σας πω ενός ισοπεδωτικού κοινού ε, τέτοιου τέλους ε, στην πολωνική οικονομία θα είναι τελείως διαφορετική από την επίπτωση στη σουηδική οικονομία και ούτω καθεξής. Και για την καινοτομία όσον αφορά την χρηματοδότηση Πρέπει να πω με κάθε σεβασμό εδώ ότι ναι, φόροι δεν είναι νέα καινοτομία. Είναι ένα από τα παλαιότερα τεχνάσματα και ένα από τα παλαιότερα δεδομένα παγκόσμια. Επίσης θα ήθελα να αποκαλύψω ένα μυστικό. Παρακαλώ λοιπόν προσδεθείτε με τις ζώνες σας, τα καθίσματά σας δεν βρίσκονται νέα χρήματα κάπου σε κάποια υπόγεια σε χρηματοκιβώτια στην Ευρώπη. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο του Ντόναλντ Ντάκα και των κινουμένων σχεδίων όπου δισεκατομμύρια κάπου βρίσκονται. Πάντα θα είναι οι πολίτες που θα πληρώνουν τους φόρους, ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει λοιπόν καινοτομία αν δεν μπορεί να βρει κανείς πολίτες να πληρώνουν φόρους κάπου αλλού για να προσθεθούν. Και στο τέλος θα πρέπει είτε μέσω υψηλότερων τιμών, είτε μέσω υψηλότερων επιτοκίων, είτε μέσω υψηλότερης φορολογίας να πληρώνουν οι πολίτες και να αρμέγονται έτσι. Μπορώ να σας ε, δώσω την ε, διασφάλιση ότι αν υπήρχε κάποια δυνατότητα θα την είχαμε ανακαλύψει με τόσα βραβεία Νόμπελ που απονέμονται σε οικονομολόγους. Όλε Σμιτ το ανέφερε σε σχέση με την ε, σουηδική εμπειρία και τις διαφορές. Θα ήθελα κάπως να διαφωνήσω μαζί του. Ήταν κάποια επιτυχία για το Λονδίνο, διότι ένα μεγάλο τμήμα των συναλλαγών από την ε, Στοχόλμη πήγε στο City του Λονδίνου και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό σε σχέση με ένα τέτοιο φόρο ε, συναλλαγών, ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών η επίπτωση για την, το κέρδος και το όφελος θα είναι υπέρ της Σανχάης εκεί θα μετατεθούν τα πράγματα και σε μια συνάντηση συζητώντας αυτά τα θέματα πρέπει να το δούμε αυτό ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών βασίζεται στην ιδέα ότι δεν είναι καλές οι χρηματοοικονομικές και συναλλαγές και πρέπει να τιμωρούνται. Εγώ έχω μια τελείως διαφορετική άποψη. Η αύξηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών τα τελευταία 30 χρόνια είναι αυτό που άλλαξε εκ βάθρων την παγκόσμια οικονομία. Αυξημένο εμπόριο, αυξημένες επενδύσεις και επενδύσεις σε χώρες όπου δεν υπήρχε το κεφάλαιο να χρηματοδοτηθούν τέτοιες επενδύσεις. Ένα χρηματοοικονομικός φόρος συναλλαγών θα είναι επιτυχής με τέτοιο τρόπο όπως αν ε, ε, επιτύχει αυτά τα οποία λένε όσοι επιχειρηματολογούν υπέρ αυτού θα είναι λιγότερες συναλλαγές, λιγότερες επενδύσεις. Δεν μπορώ να δω λοιπόν ποιο θα είναι το όφελος. Δεν θα υπάρχει όφελος για τις φτωχότερες χώρες. Δεν θα υπάρχει όφελος και κέρδος με, για χώρες με μεγάλα ελλείμματα. Διότι αγαπητοί συνάδελφοι, οι χώρες με τα μεγάλα ελλείμματα είναι εκείνες που χρειάζονται τις περισσότερες οικονομικές συναλλαγές. Και ένας φόρος επί των οικονομικών συναλλαγών θα στόχευε ακριβώς σε σχέση με αυτές τις χώρες ή τις άλλες χώρες ε, με ελλείμματα εις βάρος των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Θα είναι περισσότερο δαπανηρό, πολύ πιο δαπανηρό να χρηματοδοτούνται τα ελλείμματα. Και για αυτή την κερδοσ... την κερδοσκοπία για την οποία γίνεται λόγος, ε, κερδοσκοπία και τέτοιου είδους ε, δράσεις υπάρχουν εκεί όπου υπάρχουν ανασφάλειες και οι περισσότεροι από εμά θα ήταν ικανοποιημένοι, θα το βλέπαμε ικανοποίηση σε σχέση με την ε, ε, οικονομική κάλυψη των ε, ελλημάτων και παράδειγμα της Ελλάδας. Αλλά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό όχι κερδοσκοπώντας. Τότε θα μπορούσαμε να αυξήσουμε φορολογία έχοντας συνειδητοποιήσει ότι θα πληρώνονται αυτού του είδους τα τέλη από τους στοχότερους στον κόσμο με τα λιγότερα κεφάλαια και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο εμπόριο και περισσότερες ε, επενδύσεις ε, ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών με τα ελλείμματα. Βλέπω ότι πολύ απογοητευμένα με κοιτάζει, με μεγάλη απογοήτευση η κυρία Περβάνος Μπερές. Εν συντομία, κακή ιδέα είναι αυτή και ένα, μια τέτοια κακή ιδέα δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται πιστεύω. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της και θα ήθελα να αναφέρω ένα ή δύο σημεία. Καταρχάς η γενική αντίληψη ότι δεν υπάρχει θέμα ουδετερότητας της φορολογίας υφίσταται. Η φορολογία πάντοτε έχει επίπτωση στον ανταγωνισμό, έχει επίπτωση τα κίνητρα και στα αντικίνητρα. Δηλαδή, στην ουσία συζητάμε για αλλαγές στην φορολογία. Δεν κάνουμε αλλαγές σε μια παγιωμένη ουδέτερη κατάσταση. Αλλάζουμε τα κίνητρα και τα αντικίνητρα. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχει ένα ουδέτερο πεδίο δράσης ούτε μέσα στις χώρες ούτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της. Το θέμα είναι πώς θα μπορούσαν να, γίνουν, να υπάρξουν μοχλοί μέσα στις υπάρχουσες υποδομές. Έχουμε λοιπόν τρία θέματα. Έχουμε την επιλογή να μην κάνουμε τρίποτα Και αυτό, ε, αυτός είναι ο προβληματισμός που είναι αρκετά θεμητός. Αναρωτιέμαι εάν δεν επιβληθεί φόρος επί των πληρωμών θα μπορούσε να εισαχθεί αυτή τη στιγμή. Λόγω του ότι θα μπορούσε να αλλάξει τη δομή του φορολογικού συστήματος ή της παγκόσμιας φορολόγησης. Δεύτερον, τίθεται το θέμα ποιος δρά πρώτος. Νομίζω ότι είναι κάπως ουτοπικό να θεωρούμε ότι μετά τους G20 όλοι θα κινηθούν συντονισμένα και θα δημιουργήσουν συστήματα φορολόγησης. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώς θα μπορούσαν να κινηθούν διάφορες περιοχές και χώρες και να επηρεάσουν και τις υπόλοιπες. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα αργότερα. Το τρίτο σημείο εδώ που αφορά το ουδέτερο πεδίο δράσης είναι ότι είναι μεγάλο το άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάω για το φορολογικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ αθέμητο πεδίο δράσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα που προετάθησαν εδώ. Μου αρέσει η ιδέα ε, του φόρου συναλλαγών και το γεγονός ότι δεν ε, θεωρείται συμπληρωματικά όπως στις προτάσεις της Επιτροπής. Και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, εάν το FTT είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτός ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα στα, στα χρηματοπιστωτικά συστήματα για να υπάρξει χαμηλότερη φορολόγηση. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τη διαφάνεια. Λαμβάνω υπόψη μου το ότι υπάρχει αυτή η παγκόσμια πτυχή και ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε το πώς θα κινηθούμε. Εδώ όμω τίθεται ένα δίλημα. Δεν υπάρχει επαρκής χρόνος, αλλά ήθελα να πω ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με το αν θα μπορούσε να υπάρξει φόρος επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ε, ε, περιφερειακό και αν θα μπορούσαν να υπάρχουν περιφερειακές συμφωνίες. Με τον φόρο αυτό το όπως και με τους φόρους για το διοξίδιο του άνθρακος, το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, εταιρείε οι οποίες εγκαθίστανται κάπου και η φορολογία δεν είναι το σημαντικότερο θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον φόρο επί του διοξιδίου του άνθρακος, ε, θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάνοντας προσαρμογές στο φόρο επί του διοξιδίου του άνθρακος και να κάνουμε μια προσπάθεια συμμόρφωσης. Αυτό θα οδηγήσει μια ισορροπία αν η Ευρώπη δηλαδή κινηθεί με γοργότερους ρυθμούς σε ό,τι αφορά το θέμα της μείωσης ε, των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Είναι πολύ σημαντικό συνεπώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι καινοτομίε που έχουν σχέση με την ανάπτυξη, δεν μου αρέσουν οι εκτόσει επί των φόρων και δεν μου αρέσει το να μπαίνουν στην άκρη ε, κονδύλια που έχουν προκύψει από φόρους και μετά να αποφασίζετε το πού θα χρησιμοποιηθούν. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να ε, εξεταστούν μηχανισμοί που αφορούν τους φορολογικούς παραδείσους, τη φοροδιαφυγή και τέλος πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και τους παγκόσμιους φόρους αλλά βεβαίως αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος για την Ευρώπη. Τελευταίο σημείο. Σε κάποιο σημείο σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να θέσουμε το θέμα το πώς συμπεριλαμβάνουμε το θέμα της φορολογίας με τους δικούς μας λογιστικούς κανόνες. Αντί για το φόρο του άνθρακα θα επιθυμούσα να συζητήσουμε το θέμα της φορολόγησης των πόρων. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε φορολογώντας τους σπόρους γιατί εκεί υπάρχει ε, μεγάλη ένδυα και εκεί θα πρέπει να αυξηθεί αποτελεσματικό. Ε, Ευχαριστώ. Έχουμε ένα πρόβλημα το χρόνο αγαπητοί συνάδελφοι γιατί είναι και πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Όσο προσπαθώ να δω τι θα κάνουμε με το χρόνο, ας δώσω το λόγο στην ε, Περιβάνς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας γιατί νομίζω ότι ακόμη κι αν είναι ένα θέμα επί του οποίου αρκετοί ε, έχουν διαφορετικές ε, απόψεις, νομίζω ότι αυτό το έγγραφο είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Όταν ξεκινάμε μια συζήτηση για καινοτόμου πόρους, νομίζω ότι χρήσιμο είναι να επαληθεύουμε πάντοτε πριν γιατί τίθεται θέμα πόρων. Ίσως ε, φαίνεται μπανάλ αυτό ή περιττό, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο. πρώτη ανάγκη του φορολογικού συστήματος, της φορολογίας, είναι να εξευρεθούν πόροι για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και της αναδιανομής. Και η δεύτερη πτυχή, σε σχέση με αυτό που είπα πριν, ε, είναι η αναδιανομή, δηλαδή χρηματοδότηση της επένδυσης και των επενδύσεων και αναδιανομή. Το σύνολο των προτάσεων ε, της έκθεσης της Άννης Ποδηματά νομίζω ότι ανταποκρίνονται πλήρως στη διπλή αυτή ανησυχία που πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Σημειώνω ότι στην ευρωπαϊκή συζήτηση υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία ενίοτε ε, χρησιμοποιούνται κάπως ανεστραμμένα. Δηλαδή στο περιβαλλοντικό, στον περιβαλλοντικό τομέα. Όταν συζητήθηκε το ζήτημα των ε, ανταλλαγών ποσοστώσεων εκπομπών έγινε μια συζήτηση ακόμη και στη δική μας επιτροπή για το κατά πόσο τα καλύτερα κίνητρα για τη διόρθωση των στρεβλώσεων της αγοράς και την αποθάρρυνση της κατανάλωσης ενέργειας είναι φορολόγηση ή ένας μηχανισμός αγοράς όπως υπόθηκε με το σύστημα εμπορίας, ανταλλαγής εκπομπών. Και θεωρήθηκε ότι στον τομέα της ενέργειας, με πολύ έτσι ριζικό τρόπο εφαρμόστηκε, ο κύριος Σέκμαρκ δυστυχώς έφυγε, γιατί ήταν ένας από τους μεγάλους πέραμπους της πρότασης αυτής, της αρχής δηλαδή οριπένων ε, φορολογείται. Γιατί να μην εφαρμόσουμε ακριβώς την ίδια σύνεση και σοφία στο χρηματοπιστωτικό τομέα διότι πραγματικά υπάρχει ευθύνη των παραγόντων ε, ε, του τραπεζικού κλάδου, του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Και η ιδέα των να συνεισφέρουν αυτοί ε, σήμερα για να εξηγιανθεί, όχι μόνο να εξηγιανθούν τα δημόσια οικονομικά, αλλά για να υπάρχει δυνατότητα επενδύσεων των οικονομιών μας, μου φαίνεται μια πολύ σημαντική ιδέα που θα πρέπει να την συγκρατήσουμε. Δεύτερο επιχείρημα που ακούγεται πολύ Είμαστε σε παγκόσμιο πλαίσιο και επίπεδο και αν δεν προσέξουμε όλοι οι επενδυτές θα εγκαταλείψουν ε, την ευρωπαϊκή επικράτεια. Ο Τζόζεφ ε, Στίγκλιτς έχει πει κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα ε, και ένα από αυτά είναι ας φύγουνε, ας φύγουν αυτοί τελικά ας ε, φύγουν και θα βρούμε άλλους ε, επενδυτές στη γεραία Ήπειρο αυτή. Διότι πραγματικά παρόλα τα δράματα και τις καταστροφές είναι ένας μέρος που αξίζει και είναι ωραίο να ζει κανείς. Το να συνεχίζουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε αν δεν συμφωνεί μαζί μας ο υπόλοιπο κόσμος, μα τότε δεν πρόκειται κανείς να μετακινηθεί γιατί πάντοτε θα υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Άρα δεν θα κουνηθούμε ρούπι γιατί θα πρέπει όλοι να συμφωνούν. Με αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Αν συνεχίσουμε έτσι θα υποφέρουμε και θα αναγκαστούμε να ε, υπομείνουμε ότι θα μας επιβάλλουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα είμαστε σε αμυντική στάση εφόσον θα έχουμε απεμπολίσει την κυριαρχία μας. Τρίτο επιχείρημα που άκουσα σήμερα το πρωί και μου, έτσι, μου έκανε έκπληξη. Αυτή η ιδέα ότι η κερδοσκοπία είναι καλή και ότι τελικά οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές πάντα έχουν προσθέμενη αξία. Πρώτα απ' όλα σημειώνω ότι η κερδοσκοπία είναι ένας όρος ε, που ακόμη και αν οι οίκοι αξιολόγησης ε, που υποβάθμισαν ε, το κυρίαρχο εθνικό χρέος της Ελλάδας ε, ήρθαν στο γραφείο μου πολλοί να μου πούνε ότι αυτό το κίνημα δεν είχε κανένα κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ότι κανένας δεν αποκόμισε κέρδος οικονομικό από αυτή την κίνηση αγορές. Μα ο ορισμός τελικά της κερδοσκοπίας, τι, ποιος είναι, τι είναι η κερδοσκοπία παράγοντες της αγοράς εκμεταλλεύονται, αποφελούνται μια κατάσταση για να προσανατολίσουν τις αποφάσεις της αγοράς. Τι είναι κερδοσκοπία και τι δεν είναι κερδοσκοπία. Ε, τώρα το να αποφασίσουμε ποιο είναι το όριο ε, αυτού που κάνουμε με βάση το τι είναι κερδοσκοπία ή δεν είναι, δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα εύστοχο. Τώρα έρχομαι στην ουσία. Α, ένα τελευταίο επιχείρημα που άκουσα από την Βίκη ε, Φόρτ. ότι η έκδοση ευρωομολόγων ε, θα αυξήσει τον ηθικό κίνδυνο ε, στον προπολισμό των κρατών μελών. Μα το αντίθετο ακριβώς θα ισχύσει, κατά την άποψή μου. Αν θέλουμε να έχουμε ε, έναν λόγο στον τρόπο με τον οποίο δαπανούν τους σπόρους που εισπράττουν τα κράτη-μέλη, η έκδοση των ευρωομολόγων δίνει ένα δικαίωμα μόχλευσης. Είναι ένας μοχλός που κανένα άλλο εργαλείο δεν μπορεί να δώσει. Νομίζω λοιπόν ότι μια τέτοια προσέγγιση απέναντι στα κράτη-μέλη είναι πολύ θετική. Στην έκθεση που ψηφίσαμε για αυτή το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, στην έκθεση για την κρίση, ε, υπήρχε κάποιος ελεύθερος που ζήτησε να διαγραφεί αναφορά στο ότι θα πρέπει να είναι εφαρμοστέως αυτός ο φόρος στο ευρωπαϊκό επίπεδο αν δεν εφαρμοστεί παγκόσμια. Άρα αυτό καταψηφίστηκε. Είπαμε λοιπόν ότι αν δεν υπάρξει διεθνή συμφωνία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ως πρόδρομος, ως σκαπανέας front runner θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες ευθύνες. Φυσικά και η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά το ζήτημα της βιωσιμότητας των οικονομιών μας είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα. Και αν δεν βρούμε νέους πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τις μελλοντικές ανάγκες των οικονομιών μας, καταδικάζουμε την Ευρώπη σε ύφεση και ο κόσμος δεν μας περιμένει. Συνεχίζω να πιστεύω λοιπόν ότι με βάση τις προτάσεις της έκθεσης της Άννης Ποδηματά έχουμε πολύ σκερά στοιχεία ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να εξέλθουμε από την κρίση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο με την επιβολή κυρώσεως στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας θα ξαναδημιουργήσουμε την ικανότητα για την Ευρώπη να έχει το ρόλο της σε παγκόσμιο επίπεδο απέναντι ιδίω στη ΣΥΠΑ και την Κίνα. ιδέα λοιπόν ε, φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η ιδέα ενό φόρου άνθρακα, ώστε οι στόχοι μας οικονομικοί να ε, συνάδουν με τους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή η ιδέα επίστον των ευρωομολόγων μου φαίνονται οι ιδέες πολύ σημαντικέ. As I said... Όπως σας είπα, Έχουμε ξεπεράσει κατά 10 λεπτά το χρόνο που είχαμε προβλέψει αυτή η συζήτηση. Θα πρότεινα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και μετά να περάσουμε στο θέμα 11, γιατί ξέρω ότι οι σκιώδεις συζητητές είναι εδώ. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνουμε χωρίς διερμηνείς, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά, εάν βεβαίως συμφωνεί και όλοι Σμίτ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε χρόνο για το σημείο 11 σήμερα το απόγευμα, αλλά πολλοί από τους σκιώδεις εισηγητές ε, δεν θα είναι εδώ. Θα πρέπει να συζητήσουμε την έκθεση της κυρίας Ποδηματά που είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Θα παρακαλούσα τους επόμενους ομιλητές να καταβάλουν μια προσπάθεια να είναι όσο γίνεται πιο σύντομη για να μην μείνουμε εδώ μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Άντολιν, Μπλούμεν, Σεκλούνα, Επιτροπή, αλλά μόνο για το θέμα της αξιολόγησης των επιτόσεων. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ποδηματά και ύστερα θα περάσουμε στην έκθεση του Όλι Σμιτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγχαίρω την εισηγήτρια για την παρουσίαση της έκθεσης της ε, που έχει πολλά θετικά στοιχεία. Εντάξει, μπορώ να συνεχίσω. Και όταν κάνουμε λόγο για την Ευρώπη της καινοτομίας είναι αξιοπρόσεκτο ότι φαίνεται να κάνουμε λόγο για καινοτομία εκτός από φορολογική καινοτομία ως τμήμα επίσης για της φορολογικής ε, αυτής καινοτομίας ε, του συνόλου. Τουλάχιστον θα έπρεπε να αξίζει προβληματισμό αυτό το στοιχείο να αξίζει προβληματισμού. Πρώτον, επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο εξυγίανσης ε, δημοσιονομικής και θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ευθύνε μας Αλλά όχι μόνο για αυτό, αλλά και για πολλά διαφορετικά φαινόμενα όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, την χρηματοοικονομική κρίση και κυρίω για του στόχου μα τη ανάπτυξη, αηφόρου ανάπτυξη. Και που μας να αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας την εποπτεία και τη ρύθμιση ε, μέσα αλλά επίσης και τη φορολογία επιπλέον διότι οι εθνικές απαντήσεις είναι μη αποτελεσματικές σε πολλές περιπτώσεις και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι δεν συνεισφέρουν οι εθνικές αυτές αντιμετωπίσεις για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Τα θέματα τα οποία τίθενται επί τραπέζης είναι πάρα πολύ σκόπιμα. Η χρηματοδότηση, τα ευρωμόλογα, ο φόρος το τέλος για την έκκληση εκδιοξιδίου του άνθρακα έχουν λοιπόν αξίζουν να αντιμετωπιστούν από κοινού για τον χρηματοοικονομικό τομέα ε, φορολογικά. Και μεταξύ φορολογίας του κεφαλαίου για την εργασία που πρέπει να εξεταστεί υπάρχει επίσης μια συμμετρία μεταξύ της συνεισφοράς της βιομηχανίας όσον αφορά το φορολογικό βάρος από πλευράς φορολόγησης και που δικαιολογείται στο μέτρο που αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία. Βλέποντας όταν σημειώνονται πολύ υψηλότερα ποσοστά από την ποσοστό ανάπτυξης της οικονομίας πώς μπορεί αυτό να μην συνεισφέρει στην, ε, στον επομισμό των βαρών. Επίσης σε σχέση με την η κρίση επιπλέον καθόρισε πάρα πολύ σημαντικά βάρη για τους, ε, ε, ε, τους φορολογούμενους. Επιπλέον πρέπει να ξέρουμε ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινά κριτήρια και υπάρχει μια παγκοσμιοποιημένη ημερήσια διάταξη την αντιμετώπιση των παγκοσμιοποιημένων αυτών προκλήσεων που απαιτεί προβληματισμό και εξέταση σε σχέση με την, ε, τον φόρο, το τέλο ε, ε, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχο τη μια ή άλλη λύσης, αλλά πρέπει να προβληματιστούμε σε σχέση με αυτέ τι προτάσει, να δούμε τι μπορεί να γίνεται. Γιατί τα ευρωμόλογα. Και εδώ αυτό είναι προφανέ. και επιπλέον έχουμε ένα δυναμικό, ένα δυναμικό για την χρήση πόρων που δεν το χρησιμοποιούμε στο βέλτιστο. Αυτό είναι προφανέ. Δεύτερον, αν έχουμε συνειδητοποιήσει το θέμα τη οικονομική διακυβέρνηση, υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά όχι όλα τα στοιχεία τη οικονομική διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει μορφές ε, επιτοκίων που θα είναι επιτόκια που θα είναι κοινά. Εδώ όμως ε, έχουμε και ε, διαφορετικά συμφέροντα. Αν τα δούμε μόνο υπό το πρίσμα των κυρώσεων όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι, όταν υπάρχει μια διαδικασία για την μη τήρηση του συμφώνου, θα πρέπει επίσης να έχουμε και το θέμα της σύγκλησης των επιτοκίων και αυτό είναι σημαντικό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εξυπηρετούμε την χρηματοοικονομική ε, Ένωση. Θα, έχουμε, θα την υπονομεύουμε. Όταν, όταν έχουμε διαφορετικά επιτόκια δεν υπάρχει ένα κοινό ε, πλαίσιο κινήτρων. Και έχουμε μια συμμετρική πολιτική που θα προκαλεί προβλήματα, πιστεύω εγώ, για τη λειτουργία της ε, Χρηματοοικονομικής Ένωσης. Μετά, το τέλος του, για τις εκπομπές άνθρακα. Χρειαζόμαστε μια κοινή τοποθέτηση, αλλά επίσης επειδή έχουμε και ένα, μια κοινή εμπορική πολιτική. Καθώς έχουμε μια κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να θεσπίσουμε ποιο είναι ο τρόπο τρόπος ε, λειτουργίας ε, φορολογικά που θα πρέπει να θεσπιστεί ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα σε μια συνεκτική, συναφή πολιτική. Αυτά είναι θέματα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος και πρέπει να τύχουν σε βάθος του προβληματισμού από πλευράς μας. Ευχαριστώ. Right, it's actually uh, Leonardo because I missed him off the list, but uh, or, the. Ε, συγγνώμη κύριε Δομινίτσι γιατί τον άφησε εκτός καταλόγου. Λεωνάρδο παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ήδη ακούστηκαν πολλά. Θα ήθελα ιδιαίτερα να φερθώ στην παρέμβαση του συναδέλφου Όλη Σμιτ. Πραγματικά με εντυπωσιάζει η διάβγεια και η αναλυτική του ευφυΐα. Το θέμα που θα ήθελα να θέσω και σε εκείνον και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής είναι το εξής. Βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε γιατί κάτι συνέβη πριν από δύο χρόνια. Οι πολίτες τον χωρών μας, οι Ευρωπαίοι πολίτες, η κοινή γνώμη ζητάει από εμά απαντήσεις. Βεβαίως ορισμένες απαντήσεις τις δώσαμε ήδη, όπως για παράδειγμα το θέμα της εποπτείας. Αναρωτιέμαι όμως αν επαρκεί αυτό. Το πρόβλημα της κερδοσκοπίας υφίσταται δίχως άλλο θα πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι τρόποι λειτουργίας των αγορών και να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ τους. Σήμερα όμως δεν θα ήμασταν εδώ να συζητάμε για αυτά προβλήματα αν δεν είχε προκύψει η χρηματοοικονομική κρίση πριν από δύο χρόνια. Εάν δεν είχε παρατηθεί μια αύξηση του δημόσιου χρέου στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις, απαντήσεις που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές ακόμα και από την άποψη τη συγκράτηση των κερδοσκοπικών φαινομένων. Γιατί αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τρόπο για να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές τις ίδιε τι αγορέ. Και πιστεύω ότι αν προβληματιζόμαστε πολύ σωστά για τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και για τη ζώνη του ευρώ, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. όπως για παράδειγμα την αξιολόγηση του ευρώ. Στοιχεία που αυτή τη στιγμή επηρεάζουν σημαντικά την κατάσταση ορισμένων χωρών ε, που ενδιαφέρονται για τις εξαγωγές και που βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα υπέρογκο χρέο. Ωραία. Γκότφιν. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Uh, για τη θέσπιση αυτών με την ομάδα και είναι ότι αν φορολογείται κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν φορολογείται αλλού παγκόσμια, αυτό απλά θα μετακινηθεί σε εκείνο το τμήμα του κόσμου που δεν θα φορολογείται. Ίσως δεν σας αρέσει αυτό, αλλά αυτό θα γίνει. Φορολογείται κάτι εδώ, θα μετακινηθεί κάπου αλλού. Ρυθμίζεται κάτι εδώ, θα μετακινηθεί αλλού, ώστε να μην υφίσταται αυτών των ρυθμίσεων. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο, πρόδειλο. Και απλά και μόνο το αναφέρουμε. Το δημόσιο χρέο επίση είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε καμιά φορά σε αυτήν την ομάδα. Καμιά φορά ως είδος πολιτικής πολιτικής ε, που ακολουθείται από τους πολιτικούς. Αν ένα κράτος ε, έχει χρέος και μάλιστα βρίσκεται σε υπερχρέωση, αυτό οφείλεται στους πολιτικούς που έχουν τα ενία σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι κάτι το μαγικό ή θεϊκή βούληση και είναι κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε. Επίσης ε, για τον άνθρακα που χρησιμοποιούμε διαρκώς, άνθρακας, διοξίδιο του άνθρακα, μονοξίδιο και διοξίδιο του άνθρακα, είναι τρία διαφορετικά στοιχεία χημικά Ας μην λοιπόν αναφερόμαστε στον άνθρακα όταν δεν εννοούμε τον άνθρακα. Εννοούμε διοξίδιο του άνθρακα. Επίσης κάνουμε λόγο για την χρήση δαπάνη τεράστιων κονδυλίων για τις συναλλαγές ε, σε σχέση με τις εκκλήσεις ε, διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ είναι θέμα μόλυνσης, ε, ρήπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είμαστε ε, κάπως πιο ελαστικοί διανοητικά, πνευματικά. Ξέρουμε ότι από το 1995 είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχουμε το μικρότερο επίπεδο έκκληση ε, διοξιδίου του άνθρακα για 300 εκατομμύρια χρόνια. Επίση ξέρουμε ότι, ε, είχε, ε, ότι υπάρχει η θέρμανση του πλανήτη αλλά υπήρχε και στο παρελθόν. Ας πάψουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε ανοησίε για τι κλιματολογικέ αλλαγέ και να επιβαρυνθούν τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μα λόγω αυτή τη κατάσταση. Υπάρχει, υπάρχει η πτυχή τη κερδοφορία για κάποιους με, με αυτόν τον πανικό που δημιουργείται. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το τι γίνεται παγκόσμιο, και με, την χρηματική, και με τα, με χρηματοοικονομικά και με τα κλιματολογικά προτού πάρει τα, πράγματα, τα πράγματα τελείως στραβά. Ευχαριστώ. Um, thank you, Madam Chairman. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ. Και εγώ βρήκα ότι η έκθεση της κυρίας Ποδηματά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και έδινε πολλά ε, κίνητρα και ιδέες ε, και για την καινοτομία και την ε, καινοτόμο πλευρά σε αυτή την έκθεση. Νομίζω συμφωνώ σε σχέση με τις προτάσεις ότι η καινοτομία δεν θα έπρεπε να ερμηνεύεται σαν κάποια νέα επινοημένα χρήματα τα οποία δεν είχαμε ξανασκεφτεί στο παρελθόν διότι προέρχονται από τους ίδιους καταναλωτές αυτά τα χρήματα. Συμφωνώ σε σχέση με αυτό. Όμως η φορολογία δεν έχει σκοπό να βρει νέα χρήματα αλλά να τα διανέμει αυτά τα χρήματα. Δηλαδή στον δημόσιο τομέα, στο εθνικό ή περιφερειακό ε, επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο να παίρνουν περισσότερα κονδύλια περισσότεροι από ό,τι στο παρελθόν μέσω αυτής της διανομής. Όμως επανερχόμενοι στον καταναλωτή, στους καταναλωτές, έχει πολλές ιδιότητες ε, ο καταναλωτής και μπορεί με διαφορετικές ιδιότητες να αντιμετωπίζεται ως ε, επενδυτής ε, για παράδειγμα ή αγοραστής κάποιων προϊόντων. Κάποιες φορές είναι αγαθά, είναι καλά αυτά τα προϊόντα, άλλες φορές όχι όμως. Καμιά φορά για την φορολογία αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να δώσει κάποια μηνύματα ή να υπάρξει επιμερισμός βαρών που θα είναι δικαιότερος. Τώρα ακόμα και ως καταναλωτής ή ε, ε, παραγωγός εισοδήματος. Έχουμε και διαφορετικές κατηγορίες εισοδηματιών, ε, χαμηλού εισοδήματος, μεσαίου, μεγαλύτερου εισοδήματος, εταιρείε μικρές, μεγαλύτερες, μικρομεσαίες. Θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι για να βρεθεί ισο, ισοδίκαιος τρόπος επιμερισμού βαρών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν προτιμόμενοι τομείς που θα έχουν πλέον και προτερήματα θα πρέπει να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλοι σε μια ε, οικονομία. Το ίδιο και για τις οικονομικές δραστηριότητες. Υπάρχει κακή ε, τέτοια παραγωγή, τότε αν ρηπαίνεται η ατμόσφαιρα να πληρώνει ο ρηπαίνων. Να πληρώνεται, να, να καταβάλει χρήματα, διότι θα πρέπει να αποτρέπουμε, να αποθαρρύνουμε τέτοιου είδους ε, δράσεις που δεν είναι επωφελείς για την κοινωνία. Ενθαρρύνω λοιπόν το να είμαστε καινοτόμοι, να βρούμε τρόπους για τον επιμερισμό βαρών και να βρούμε τρόπο να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα διότι όπως γνωρίζουμε υπάρχει μετάθεση φορολογικών βαρών, tax shifting και εκείνοι που πληρώνουν αυτούς τους φόρους θα πρέπει να δούμε αν θα είναι η τελική ε, ε, υπεύθυνη της ε, φορολογίας για τον επιμερισμό των βαρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τώρα στην Επιτροπή γιατί πολλοί αναφέρθηκαν στην αξιολόγηση επιπτώσεων. Η Επιτροπή λοιπόν. Θερμή παράκληση να είστε σύντομοι γιατί πραγματικά πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να κάνει μια έκθεση αξιολόγησης μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό αναφέρεται σαφώς στην ανακοίνωση της 7ης Οκτωβρίου και θα πρέπει να πω ότι από την άποψη της Επιτροπής λυπούμε αυτά για τις αναφορές που έκανε η συγγήτρια σχετικά με την αδυναμία μας να αντιδράσουμε. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο που θα πρέπει να συζητηθεί στην αξιολόγηση επιπτώσεων και η συζήτηση το κατέστησε απόλυτα σαφές. Ένα σημείο. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον στόχο του φόρου επιχειρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μιλάμε για ένα φάσμα διαφορετικών φόρων και αυτό οδηγεί στη δημιουργία σύγχυσης όχι μόνο στα πλαίσια αυτής τη συζήτησης αλλά και εκτός. Άκουσα σαφώ την αναφορά στην έλλειψη καινοτομιών από πλευρά τη Επιτροπή. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή υπήρξε καινοτόμο στην ανακοίνωσή τη και αναφέρθηκε στο φόρο επιχειρηματοπιστωτικών ε, δραστηριοτήτων. Αυτό αφορά τα εισοδήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Δίχω άλλο πιστεύουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τομέα για διερεύνηση και μπορεί να αποτελέσει και ένα σημείο αναφορά για την εξέταση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι χρηματοπιστωτικοί φόροι. Τέλο, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά ε, στο εύρο των φόρων αυτών. Πολλές ε, συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά με το θέμα του, φόρου, ε, του τέλους χαρτοσύμου. Το τέλος ε, χαρτοσύμου ε, είναι ένα πολύ πολύπλοκο εργαλείο. Είναι όπως τα παράγωγα. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε τα παράγωγα θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε χωρίς να πλήξουμε το εμπόριο. Δεν είναι σαφές αυτό. Θα πρέπει είτε να εντοπίσουμε τι είναι ζημιογόνο και τι δεν είναι όπως αναφέρθηκε Βεβαίω ε, ο βραχυπρόθεσμος ορισμό δεν είναι ε, δεκτός. Το θέμα είναι να δούμε αν η ζημιογόνος δράση συνεχίζεται και θα πρέπει όμως να δούμε κατά πόσον και το καλό και το κακό συμπορεύονται. Η αξιολόγηση επιπτώσεων θα πρέπει να εξετάσει αυτές τις πτυχές από κοντά και τελικά, τελευταίο σημείο, στην Επιτροπή έχουμε απόλυτη συνείδηση της ανάγκης να υπάρξει μια γενική άποψη των επιπτώσεων που θα προκύψουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στην Άννη πάρα πάρα πολύ σύντομα γιατί η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα εκτενής και θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε όταν περάσουμε στην επόμενη ανταλλαγή απόψε χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Okay. Okay. Ε, όσο πιο σύντομα ε, γίνεται, ξεκινώντα από την τελευταία παρατήρηση εκ τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, ε, νομίζω ότι στην έκθεση αλλά και στην παρουσίαση που έκανα πριν δεν είπα τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, το γεγονό δηλαδή ότι έχει μεσολαβήσει πολλή χρόνο. Ε, για να ε, υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που εδώ και ένα χρόνο ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή την εκπώνηση μιας μελέτης επιπτώσεων ε, που ανακοινώσατε μόλις ότι θα την υποβάλλετε το καλοκαίρι. Με αφορμή αυτό, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, γιατί είναι ένα θέμα που ετέθη από διάφορους συλλαδέρφους, ότι σε αυτό, για να ξεκινήσω από αυτά στα οποία συμφωνούμε, μελέτη επιπτώσεων, είναι προφανές ότι όλοι συμφωνούμε ότι ε, είτε υποστηρίζουμε τη θέσπιση ενός φόρου από των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε όχι όλοι συμφωνούμε ε, ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια μελέτη επιπτώσεων που να ε, συνυπολογίζει να λαμβάνει υπόψη τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. ένα δεύτερο σημείο στο οποίο επίσης συμφωνούμε είναι προφανές ότι είναι καλύτερα για όλους το ευκταίο το επιδιωκόμενο είναι να πάμε σε μια παγκόσμια συμφωνία να εφαρμοστεί ένας τέτοιος φόρος σε παγκόσμιο επίπεδο όπως νομίζω ότι ε, με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με το χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τότε που έχει ανοίξει η συζήτηση για, την ανάγκη θέσπισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι η στιγμή να δούμε πώς πώς δηλαδή είναι, ε, ποιος είναι ο καταλληλότερος, ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να φτάσουμε στην επίτευξη μιας παγκόσμιας ε, συμφωνίας. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πιέσει περισσότερο αποτελεσματικά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο, διότι υπήρξαν αρκετοί συνάδελφοι που μίλησαν για τους κινδύνους να πληγεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, να φύγουν οι δραστηριότητες αυτού του τύπου οι συναλλαγές εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας ότι εάν είχαμε αυτήν την ε, λογική και πριν από τρία χρόνια όταν συζητάγαμε για το κλιματικό ενεργειακό πακέτο ε, και υπήρχαν και τότε πολύ ισχυρά επιχειρήματα ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα υποστεί μεγάλο πλήγμα ότι θα υπάρξει αυτό που ονομάσαμε διαφυγή ε, άνθρακα ακριβώς για να οδηγήσουν στην μη ανάληψη δεσμευτικών στόχων ε, σε σχέση με την ε, αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Και καταφέραμε το 2008 και ευτυχώς και προχωρήσαμε μονομερός, μόνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών, για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων. Και δεν υπέστη κανένα πλήγμα, ίσα ίσα ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από τη συμφωνία αυτή και το δεύτερο είναι ότι εάν δεν είχε φτάσει η ευρωπαϊκή ένωση σε αυτή τη συμφωνία μόνομερώς ε, πολλές χώρες που μονομερώς επίσης στη συνέχεια προχώρησαν ε, στη θέσπιση δικών τους στόχων για τη μείωση των εκπομπών παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να φτάσουμε σε παγκόσμια συμφωνία. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη γνώμη μου, το γεγονός δηλαδή ότι μπήκαμε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια έπαιξε καταλυτικό ε, καταλητικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Ε, ένα άλλο σημείο ευθύνεται ή δεν ευθύνεται ο χρηματοπιστωτικό τομέα για την κρίση. Όλοι νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει αυτή τη συζήτηση στο πλαίσιο και τη συζήτηση τη έκθεση ε, ε Μπέρε. Επιμένω ότι υπάρχει κοινό τόπο επ' αυτού. Ε, νομίζω όμως ότι ε, επειδή όλοι, όλοι <laughs> νομίζω ότι ε, επειδή ε, υπήρξε μια αναφορά ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, πολιτικοί, υπουργοί από διάφορες χώρες, τι έχουμε κάνει εμείς, ποια είναι η δική μας συμβολή σε αυτή την κρίση και επειδή πιστεύω ότι αυτό ενδεχομένως συνδέεται, μάλλον συνδέεται με την ελληνική κρίση, ε, με, με την κρίση χρέους που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μου, θέλω να πω ότι, ε, να επαναλάβω ότι η κρίση για την κρίση του 2008 δεν νομίζω ότι υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι ευθύνεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Από εκεί και μετά έχουμε πει και έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι για τη διάχυση της κρίσης αυτής για τη μετατροπή της σε κρίση χρέους υπάρχουν ευθύνες εθνικές και ευρωπαϊκές ευθύνες στην οικονομική διακυβέρνηση στο οικονομικό στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι ε, μας αφορά είναι απολύτως γνωστό και δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση ότι τις έχουμε αναλάβει πλήρως και έχουμε αναλάβει και το κόστος αυτών των εσφαλμένων επιλογών του παρελθόντος. Από εκεί και μετά όμως συζητώντας για, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τους τρόπους συμβολής στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, που είναι πέρα πάσης αμφιβολίας ένα πρόβλημα της Ευρωζώνης και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε στην εθνική διάσταση σε καμία περίπτωση. Συμφωνώ με τον Σβέν επίσης ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ιδεολογικοποιήσουμε ε, αυτή τη συζήτηση. Πρέπει όμως, και αυτό το πιστεύω και το υπογραμμίζω, ε, αυτή τη συζήτηση όλοι μας να καταβάλουμε μια προσπάθεια να την ευρωπαϊκοποιήσουμε έστω και αν ε, ο όρος είναι ενδεχομένως κάπως δηλαδή η επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων αφενός και αφετέρου η μεγάλη συζήτηση το είπαν διάφοροι συνάδελφοι ότι δεν είναι λογικό να συζητάμε για νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς να είναι σαφές με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουμε τους πόρους, τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτά τα νέα καινοτόμα εργαλεία. Βασικός γνώμονας ε, και στις δύο περιπτώσεις είναι κατά τη γνώμη μου ε, ε, το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Ευρωομόλογα, έχει δίκιο η κυρία Χούμπνερ, άλλο πράγμα τα ευρωομόλογα για τη χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών σχεδίων, άλλο πράγμα τα ευρωομόλογα για την κοινή διαχείριση χρέους επί του παρόντος χρησιμοποιείται ο όρος ευρωομόλογα και για τις δύο περιπτώσεις αλλά θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να διακρίνουμε ε, αυτά τα δύο πράγματα διότι ε, είναι διαφορετική η λογική τους και εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους. Σε ό,τι αφορά τα ευρωομόλογα για την κοινή διαχείριση χρέους που είναι ένα ζήτημα που ετέθη από διάφορους συναδέλφους σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει υπονομευτικά ε, στη μεγάλη συζήτηση ε, που βρίσκεται σε εξέλιξη ε, για την οικονομική διακυβέρνηση και για την θέσπιση κυρώσεων απέναντι στα κράτη μέλη που θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέους. νομίζω ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο και να εξισορροπήσουν αυτή τη συζήτηση γιατί ακριβώς η ευρωπαϊκή ένωση δεν λειτουργήσε μέχρι σήμερα στη λογική μόνον του μαστιγίου λειτουργήσε και προχώρησε στη λογική ενός συνδυασμού ε, μαστιγίου και καρότου. Ε, έχω και άλλα πράγματα να πω ασφαλώς γιατί υπήρξαν πάρα πολλέ παρατηρήσεις. Σέβομαι Σάρων το γεγονός ότι ε, είναι πολύ προχωρημένη ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προτάσεις σας και τις παρατηρήσεις σας και φαντάζομαι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και τις επόμενες εβδομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννη. Το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, αρχική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα ήταν η 12η Νοεμβρίου. Πιστεύουμε όμω, ε, και υπήρξε και σχετικό αίτημα, ότι καλό θα ήταν να παραταθεί. Συμφωνεί η συγγήτρια. Και από τεχνική πλευρά είναι εφικτό αυτό. 16 Νοεμβρίου, λοιπόν, λίγη προθεσμία. Την επόμενη Τρίτη δηλαδή. 12 το μεσημέρι. 16 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. 30 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, δεύτερη φορά θα τις εξετάσουμε στις 24, μάλλον 13, μετά 24 και 23 Ιανουαρίου και Φεβρουάριος δεύτερη Ολομέλεια. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ και λυπούμε γιατί τώρα κάπως συρρυκνώνουμε ένα θέμα πάρα πολύ επίσης ενδιαφέρον για τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών δηλαδή. Πέντε λεπτά θα έχουμε ακόμη υπηρεσίες διερμηνίας και μετά θα περάσουμε στα αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ σημαντική και η συζήτηση που προηγήθηκε. Όλες σα ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να πω επίση θα έπρεπε ήδη να έχω πάει κάπου αλλού. Θα δώσω στον Έντουαρτ Τσικλούνα την Προεδρία. No, I don't need to be somewhere else. Εγώ δεν χρειάζεται να πάω κάπου αλλού. Και θα με ανεχτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Για Όπως είπε η πρόεδρος, πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική οδηγία. Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να γίνει μια συνάντηση μεταξύ των σχεδόν εισηγητών την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα. Έχετε δει το έγγραφο εργασίας. Είδατε ότι είναι ένα πλαίσιο βάσει το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Και νομίζω, νομίζω ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι. Η παλιά οδηγία υφίσταται εδώ και 10 χρόνια, όπως γνωρίζετε, και υπάρχει ανάγκη για καλύτερη προστασία των επενδυτών και για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο. Θα έλεγα, εν συντομία, ότι η οδηγία αφορά την καλύτερη κάλυψη θα περάσουμε από 20 σε 50.000 ευρώ κάλυψη από ε, αποπληρωμή το αργότερο με 5 μήνες μετά βελτιωμένη ενημέρωση περισσότερες σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο είναι καλυμμένο το ενεργητικό τους μακροχρόνια και η υπεύθυνη χρηματοδότηση θα υπάρξει μια προχρηματοδότηση. Η Επιτροπή προτείνει ένα μηχανισμό δανεισμού μέσα από εθνικά προγράμματα, μια ευρύτερη προστασία. Θα πρέπει να προστατεύονται οι επενδυτές και θα πρέπει να προφυλάσσονται από την πτώχευση τρίτων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, επενδυτικό ταμείο. Υπάρχουν Αγαπητοί συνάδελφοι, τρία βασικά θέματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας αυτά ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής καταρχάς, η κάλυψη των προγραμμάτων αυτών προτείνεται να επεκταθεί και σε επιχειρήσεις που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε οποιαδήποτε επενδυτική επιχείρηση. Υπάρχουν ε, επιχειρήματα που αφορά την επέκταση της ε, του στόχου αυτού. Οι καταναλωτές προστατεύονται σήμερα από τις διάφορες διατάξεις. Για παράδειγμα υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας Το ευρύτερο αυτό επίπεδο σημαίνει ότι χρειάζονται νέες μέθοδοι για να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Το ευρωπαϊκό Ταμείο, το ΕΦΑΜΑ, υπολόγισε ότι το προτινόμενο επίπεδο θα χρειαστεί μια συμβολή περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ που δυνητικά τελικά ε, θα καλύψουν ένα διάστημα 10 ετών. Δύο, οι αρχέ του μηχανισμού χρηματοδότηση. Η Επιτροπή προτείνει όλε οι χώρε μέλη να δημιουργήσουν ένα απόθεμα εν ώψη των μελλοντικών ζημιών. Θα πρέπει να είναι το 0,5% τη αξία του ενεργητικού που καλύπτεται από την προστασία του προγράμματο και θα πρέπει να χρηματοδοτείται με συνεισφορέ από τι χώρε μέλη και από επενδυτικά ταμεία. Υπάρχουν ε, ε, επιχειρήματα υπέρ και κατά για έναν εναρμοσμένο τρόπο χρηματοδότηση σε όλες τις ευρωπαϊκές ε, χώρες. Σήμερα έχουμε 29 με συγχωρείτε, 39 διαφορετικά προγράμματα επενδύσεων στις διάφορες χώρες μέλη. Ε, με προγράμματα αποζημίωσης των επενδυτών. Ενδεχομένω δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε λαμβάνοντα υπόψη ε, του κίνδυνου. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, δημιουργίας απολών ταμείων που θα αυξήσουν το κόστο και τη διοίκηση ε, αυτού του συστήματο. Το επίπεδο των αποζημιώσεων. Η Επιτροπή προτείνει ένα υψηλό επίπεδο ελάχιστη αποζημίωση, δηλαδή 50.000 αντί για 20.000. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια σημαντική αύξηση των αποζημιώσεων δηλαδή 150% σε σχέση με, με το τρέχον επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις πληρώθηκαν μικρά ποσά. Η υψηλότερη κάλυψη θα μπορούσε να έχει χαμηλότερη προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των επενδυτών. Κατά την άποψή μου αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω και θα επιθυμούσα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Υπάρχει ανάγκη για μια δελεχέστερη ανάλυση και συζήτηση των προτινόμενων αλλαγών σε ό,τι αφορά τα τρία αυτά τα θέματα. Θα επιθυμούσα να εστιάσω την προσοχή μου στι προτάσει αυτέ τη Επιτροπή που, κατά την άποψή μου, την κάνουν τη υποστήριξη των μελών και ελπίζω έχουν την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπαμε την πρόταση τη ε, ευθυγράμμιση ε, ε, των διευκρινήσεων και την πρόληψη για τη μερική αποσμίωση και καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών. Ανακεφαλαιώνοντα, συνεπώ, προτείνω ένα fast track για την εφαρμογή των, της οδηγίας. Το, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει, γιατί θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη, ενδεχομένω δεν θα πρέπει να επεκταθεί και στους χρήσεις. Γνωρίζουμε ότι οι χώρε μέλη προβληματίζονται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Το επίπεδο χρηματοδότησης θα μπορούσε επίσης να συζητηθεί. Το κόστος προχρηματοδότησης είναι επίσης ένα θέμα προβληματισμού, εναλλακτικές ε, πηγές δανεισμού θα πρέπει να διευκρινιστούν. Κατά συνέπεια και συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω μάλλον τολμήσω να πω, ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα πιο light, σε ένα πιο ελαφρύ καθεστώς έτσι ώστε να περάσει με πιο ταχύ ρυθμό μέσα από αυτέ τι διαδικασίες. Δεν είμαι τόσο πολύ υπέρ τη πρώτη ανάγνωση. Νομίζω ότι έγιναν πάρα πολλέ πρώτε αναγνώσει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και δεύτερες και τρίτες και τώρα προσπαθούμε να το αντισταθμίσουμε αυτό με αυτούς ε, τους ε, τριμερείς ε, διαλόγους. Έχω κάποιο σκεπτικισμό για αυτό το θέμα. Μήπως θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία και μια ευρεία συνένεση. Εγώ θα προτιμούσα μια πρώτη ανάγνωση και αυτό θα ήταν υπέρ και των καταναλωτών και των χωρών μελών και των ε, ε, τραπεζών και των επενδυτικών εταιριών. Ευχαριστώ όλοι Σμιτ. Παίρναμε στους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας χαροποιήσει ιδιαίτερα αυτή η πρόταση Στόχος είναι να αυξηθεί η προστασία των επενδυτών. Αυτό είναι ένα σύστημα που απεδείχθη ότι είναι αρκετά εξισορροπημένο από την άλλη πλευρά. Η νέα πρόταση δεν θα πρέπει να επιφέρει ένα επιπλέον άχθος. Νομίζω ότι θα μας πληρώσουν στη τελευταία ανάλυση οι επενδυτές. Θα ήθελα να αναλύσω τα διάφορα θέματα που έθεσε ο συνάδελφος. Η πρόταση της Επιτροπής ευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στον τομέα των usage. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά μην ξεχνώντας ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους επενδυτές, οι οποίοι είναι εντελώς ακάλυπτοι. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο της αποζημίωσης, και το ότι περνάει από 50 στις 20.000 ευρώ είμαστε υπέρ γιατί κατά την άποψή μας θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό το θέμα και να έχουμε κατά νου τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των επενδυτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της εναρμόνισης θα πρέπει να ε, προταθεί μια πλήρης εναρμόνιση. Αυτή είναι μια άποψη που μας βρίσκει σύμφωνους. Εγώ πιστεύω ότι η πρόταση αυτή είναι δυνατή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περιπτώσεις ανάγκης μπορεί να υπάρξει μια κάλυψη με εισφορές εξπόσεις. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες σε αυτό το τομέα εμεί είμαστε υπέρ μια εναρμόνιση. Μπορώ ότι πιστεύουμε ότι απαιτείται ένα επίπεδο ελαστικότητα για να υπάρξει προσαρμογή στι ανάγκε των ε, χωρών μελών. Σε κάθε περίπτωση το θέμα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί εκτενώς στι επόμενε συζητήσει μας. Τέλος, σε ό,τι ε, αφορά τις χώρες μέλη υπάρχει μια υποχρέωση που ορίζεται από την Επιτροπή. Τα μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τα συστήματα αυτά προστασίας και θα επιθυμούσα να υπάρξει ένα σύστημα που να βασίζεται σε εθελοντική βάση και όχι σε υποχρεωτική βάση. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ τελειώνει η διερμηνία. Σας ευχαριστούμε. Next